Παρακαλώ όλες και όλοι να καθίσετε και ο ίδιος ο εισηγητής, παρακαλώ. Ρωτώ και αν έχετε τις ε, κάρτες σας για τις ε, ψηφοφορίες. Μία, μία ψηφοφορία προβλέπεται σήμερα για τα ελαφρά οχήματα, ελαφρά εμπορικά οχήματα και θα ακολουθήσει το υπαριθμόν 10 για θέματα ε, βιωσιμότητας ε, και της εκβιομηχάνησης της Ευρώπης, παραγωγή της ανταγωνιστικότητας κλπ. Και μετά έχουμε την συνάντηση με τον Επίτροπο κ. Μπόρζ. Θα αρχίσουμε με την ενοποιημένη 1. Μια στιγμή. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, Consolidated 1, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην ενοποιημένη 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Μετά τραν 11 υπέρ, κατά. Ένα λεπτό δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία TRAN 11. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 3 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ομοίως 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 και τραν 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τραν 14 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία μεταφορών 14, τραν 14, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τέλος, εγκρίνεται. δύο. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τρία. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε εννέα. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην Ήτρε 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 με την Τραν 16 μαζί υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 81 και την τραν 16. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 82 και τραν 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και προχωρούμε με ένα άλμα στην 11 συν ήτρα 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί η 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 14 ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται ήτρε 1 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Ήτρε 1 ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται προχωρώ με ένα άλμα στην 18 και τραν 2 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 συν τραν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έρχομαι στην 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ακολουθεί η 30 συν τραν 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Και ακολουθεί η υπαριθμόν 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Ακολουθεί, ακολουθεί η τραν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, επαλήθευση, επαλήθευση. Την 39 του κυρίου Φλόρεντς. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Και συνεχίζουμε με την 44. Τραν 9 λοιπόν, γιατί απορρίπτεται, έχει απορριφθεί μόνο 44. Υπέρ, τραν 9, κατά, τραν 9, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τραν 9. Ψηφίσατε, τέλος. εγκρίνεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρώτη τελική ψηφοφορία αρχίζει. Ηλεκτρονικά βεβαίως. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος της ψήφου. 45 υπέρ 3 κατά 8 αποχές. Τελική ψηφοφορία τώρα για το νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα. Επίσης ηλεκτρονικά αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 53 υπέρ μία, 4 ε, μάλλον κατά και μία αποχή. Και τώρα θα ρωτήσω τον εισηγητή. Επιθυμείτε να αρχίσετε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, ναι ή όχι. Παρακαλώ την Επιτροπή, την παρούσα Επιτροπή, να μου χορηγήσει την διαπραγματευτική εντολή. Ναι, ο Χόλγερ Κράμερ λοιπόν θέλει, αλλά πρέπει να το επανεξετάσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και χρειάζεται να ταχθούν τουλάχιστον 35 συνάδελφοι υπέρ της χορηγήσεως της εντολής. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Σαφέστατα εγκρίνεται η χορήγηση της εντολής. Συγχαρητήρια και απευθύνω το καλό ορίσατε στην ομάδα επισκεπτών της συναδέλφου μου από το Βερολίνο. Εγώ για μια στιγμή είχα την αίσθηση ότι το μισό Βερολίνο είχε έλθει εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν, θερμό καλώς ορίσατε και μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις συζητήσεις μας. Όσοι τώρα από τους συναδέλφους επιθυμούν να παραμείνουν πολύ ευχαρίστως, όσοι επιθυμούν ή έχουν άλλα σχέδια, να εγκαταλείψουν την αίθουσα ήσυχα και αθόρυβα. Συνεχίζουμε τώρα με την νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Με εισηγητή τον κύριο Σιμάνσκι που θα τον παρακαλέσω ευθύς αμέσως να λάβει το λόγο. Ωστόσο παρακαλώ όλες και όλους να διακόψτε τις συζητήσεις ώστε να μπορέσει ο συνάδελφός μας να λάβει τον λόγο μέσα σε κλίμα ευπρέπειας. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης και η δική μας Επιτροπή γνωμοδοτεί όπως πολλές άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε ε, με αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή την Επιτροπή Βιομηχανίας. Έχετε λάβει το σχέδιο της νομοδότησής μου. αποστολή μου ήταν να ε, τονίσω το ρόλο της βιομηχανίας στην Ευρώπη που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης αλλά και τις διατηρεί. Είναι βασικό στοιχείο στην ε, στρατηγική μας για την απασχόληση και την ε, πλήρη απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είμαι πλήρως πεπισμένος και βαθύτατα ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για να ε, βοηθήσει τη βιομηχανία και να τη σώσει ε, μπορεί να είναι ισόρροπη. Τι εννοώ, από τη μια μπορούν να υποστηριχθούν οι βιομηχανίες ε, για να διατηρηθούν στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων. Από την άλλη όμως θα μπορούσε η στρατηγική αυτή να έχει ως εξή. Να περιορίζει οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ε, στο περιβάλλον. Βέβαια θα μου πείτε αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου. Ε, γίνεται εάν ε, συνεργαστούν σωστά και συντονιστούν όλα τα ενεχόμενα μέρη. Εγώ πιστεύω ότι μια βιώσιμη βιομηχανική πολιτική μπορεί να εφαρμόζεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε και μια κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική. Αν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ηγέτης στον αγώνα και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και το τίμημα που καλούνται να καταβάλουν ε, οι βιομηχανίες μας. Τώρα βλέπουμε να φεύγουν ε, βιομηχανίες που παράγουν πολύ διοξίδιο του άνθρακα και να μεταγκαθίστανται. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει σαφή διάκριση, μάλλον να φέρει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στην ε, τιμολόγηση της ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι προτείνω εγώ λοιπόν. να βρούμε πιο φθηνές ε, πηγές, μορφές παραγωγής ενέργειας, μη συμβατικές, παράδειγμα το σκιστολιθικό αέριο. Και η διαφυγή της βιομηχανίας που παράγει πολύ διοξίδιο του άνθρακα, ε, τελικά είναι κατά της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας στην Ευρώπη ε, δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Διότι είναι μικρός ο αντίκτυπος, ε, η ρήπαση του περιβάλλοντος ε, από διαδικασίες παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου και σε σχέση με κλάδους της βιομηχανίας που καταναλώνουν ε, πολύ ενέργεια, οι λεγόμενες ενεργοβόρες. Έχουν μειωθεί οι εκπομπές ρήπων και συγκεκριμένα διοξιδίου του άνθρακα πρόσφατα κατά 8% με νέες τεχνολογίες, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε αυτές ε, τις μορφές ενέργειας ε, χρειαζόμαστε ε, υλικά που έχουν παραχθεί από ενεργοβόρες βιομηχανίες, ας πούμε ένα συγκεκριμένο είδος ε, γυαλιού. Ε, παρακαλώ να σκεφτούμε και τις προθεσμίες, λίγη στις 15 του μηνός Μαΐου η προθεσμία και παρακαλώ να παραμείνουμε σε επαφή για να καταλήξουμε για την γνωμοδότησή μας. Ορισμένοι θεωρούν ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ είναι το άσυλο της ε, περιβαλλοντικής προστασίας. καλούμαστε όμως να συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές, προκειμένου με την Επιτροπή Βιομηχανίας Ενέργειας κτλ. Ευχαριστώ. das äh, Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ε, αυτό είναι αμφισβήτητο, δεν το αμφισβήτη κανείς. Ε, εκτός από τους ε, έχω άλλους τρεις συναδέλφους και την κυρία Κάντενμπαχ, δεν ξέρω αν ξέχασα ο κύριο Παναγιώτοφ, μα εσείς είστε σκιώδης. Μην ζητάτε το λόγο σκιώδης, σα ξέρω. Ε, σας έχω λάβει υπόψη μου. Ποιος ε, θα μιλήσει πρώτος? Ε, ε, ο κύριος Λάινεν εκπροσωπεί τη Γιούντιτ Μέρκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο που ε, έγραψε τη γνωμοδότηση, τον κύριο Σιμάνσκι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, σε πολλές παραγράφους. Αυτά που αναφέρονται είναι ακριβώς τα αντίθετα από εκείνα που επί σειρά ετών έχουμε εμείς εκπονήσει και αποφασίσει. Προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι για μας ε, κινητήρια δύναμη για την ε, επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης και προοπτική για το μέλλον, για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας. Και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ούτε τροχοπέδι, ούτε αρνητικό παράγοντα όπως αναφέρει η γνωμοδότηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι Ε, το μέλλον στην Ευρώπη ε, ε, σημαίνει οικονομία στη διαχείριση των πόρων που φθήνουν και χρειάζεται νέα οικονομία, νέες επενδύσεις. Μέρη έχει γίνει αυτό ήδη. Προσωπικά θεωρώ ότι η γνωμοδότηση αυτή χρειάζεται πολλές τροπολογίες και επεξεργασία για να έχει πιο ευνοϊκή ε, προβολή και βάση η προστασία του περιβάλλοντος και οι ανανεώσιμες ε, και βιώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως στη μεταβατική περίοδο υπάρχει και ένα κόστος και αντίστοιχα θα κινηθούν και τα τιμολόγια και ο ανταγωνισμός ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με άλλους παγκόσμιους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Παρ' όλα αυτά, μια στρατηγική για το μέλλον δεν μπορεί να συνίσταται στο να τερματιστούν τώρα όλα τα μέσα προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Όχι, θα πρέπει να βρεθεί το σωστό εκείνο πλαίσιο ή το σωστό μέσο για να ε, αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις που είναι πραγματικά εκατομμυρίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτοφ, παρακαλώ. Φιλελεύθερη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι η επαβιομηχάνηση της Ευρώπης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη. Βέβαια θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο με μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον, με πράσινες τεχνολογίες. Όσον αφορά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, νομίζω ότι ε, η συζήτηση αυτή θα μας απασχολήσει πάρα πολύ πριν την επόμενη ψηφοφορία που θα έχουμε, προκειμένου να επιλύσουμε τα εκκρεμία ακόμα ζητήματα που έχουμε. Όσον αφορά τώρα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή προφανώς εξαρτάται από την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης, καθώς επίσης όμως και από τα καλύτερα βιωτικά επίπεδα στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, να προχωρήσουμε με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. Ευχαριστώ. Από τους Πρεσίνους ο κύριος Μπάς Έκχοτ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συντάκτη της γνωμοδότησης για τις νοθεσίες αυτές που μας δίνει και τη γνωμοδότησή του. Δεν θα σας κάνει εντύπωση το ότι δεν συμφωνώ απολύτως με τα όσα έχουν καταγραφεί στη γνωμοδότηση αυτή και προφανώς θα περιμένετε κάποιες τροπολογίες στη γνωμοδότησή σας τροπολογίες οι οποίες διαφέρουν πάρα πολύ τελικά από το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να στείλει ο εισηγητής με την έκθεσή του. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το πραγματικό μέλλον της Ευρώπης και νομίζω ότι όλοι στην αίθουσα αυτή συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε προφανώς μια βιομηχανία στα πλαίσια της Ευρώπης. Το μεγάλο όμως ερώτημα είναι το ακόλουθο. Τι είδους βιομηχανία θέλουμε στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πιστεύω. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία της Ευρώπης με μια κοινωνία που όλο γυράσκει και ανοιγόμενη περισσότερο προς τον έξω κόσμο και προς την γενικότερη ανταγωνιστικότητα, ξέρετε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν με μια γυράσκουσα κοινωνία. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα είναι χαμηλότερη από τις συναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ινδία. Και ως προς αυτό, λοιπόν, εμείς θα μειονεκτούμε. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει, βέβαια, η προοπτική αυτή. Επίσης είμαστε μια περιοχή η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από ενεργειακούς πόρους, υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε αρκετούς φυσικούς πόρους, επομένως καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε μια ευάλωτη κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που θα μας καταστήσουν ανταγωνιστικούς ε, παγκοσμίους. Θεωρώ όμω ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αν επενδύσουμε στην κοινοτομία. Μέσω τη κοινοτομία η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Δεν θα το καταφέρουμε αυτό με του φυσικού μα πόρου ή με την γυράσκουσα κοινωνία μα κ.ο.κ. Επίση, στη γνωμοδότηση αυτή βλέπουμε ότι υπάρχουν 7 μονοσημεία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε με κάποια από τα σημεία τα οποία δεν αληθεύουν τελικά. Α δούμε τι υψηλέ τιμέ ενέργεια, μα είναι υψηλέ οι τιμέ στην ενέργεια εξαιτία τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείξτε μου μια μελέτη η οποία πραγματικά να καταδεικνύει ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι κινούν τι τιμέ τόσο ψηλά θέσουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση εδώ, ας δώσουμε πραγματικά στοιχεία. Αυτό το οποίο θα προτείνω εγώ είναι να δούμε καταρχάς ποια είναι τα δυνατά σημεία της Ευρώπης για το μέλλον, η καινοτομία προφανώς, και τι είδους καινοτομία θέλουμε σε ποιου τομεί θέλουμε πραγματικά να βρεθεί η Ευρώπη στην ηγετική θέση. Θέλουμε μια καινοτομία η οποία θα οδηγήσει σε χαμηλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ω προ αυτό μπορούμε να είμαστε παγκοσμίω ανταγωνιστικοί. Και έπειτα πρέπει να δούμε συγκεκριμένου τομεί, όπω τον τομέα τη χαλιβουργία. Αν δείτε την υπερπαραγωγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτό, θα δείτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι έχουμε τον οικοδομικό τομέα, καθώς επίσης και το τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που δεν θα καταφέρουν να ανακάμψουν όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ε, πρώτερα επίπεδά τους, αυτά δηλαδή που είχαν το 2006-2007. Στο μέλλον δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση όσον αφορά τις οικοδομές ή τα αυτοκίνητα. Θεωρώ ότι εκεί πέρα που υπάρχει πραγματικά μεγάλη ζήτηση όσον αφορά το τομέα της χαλιβουργίας είναι ο τομέας της ολικής ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία να κινηθεί περισσότερο προς το τομέα αυτό της ολικής ενέργειας. Θα πρέπει δηλαδή να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τομείς μεταξύ τους. Εκεί υπάρχει προσφορά και υπάρχει ζήτηση. Και θα δείτε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το μόνο τρόπο τελικά για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Επίσης πρέπει να δούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την λεγόμενη βιοοικονομία μέσω του χημικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές, αλλά πρέπει να καταφέρουμε να κοινοτομήσουμε ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί διαφορετικά θα μείνουμε πίσω. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε και κάποιες ε, πολιτικές για τις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να βοηθούν όμως την κοινοτομία. Γι' αυτό και εμείς ως πράσινοι προωθούμε τις πολιτικές για τις κλιματικές αλλαγές, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης, η οποία πρέπει να γίνει με τρόπο οικολογικό, με τρόπο πράσινο. και αυτό ακριβώς θα συμπεριλάβουμε στις ε, τροπολογίες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τροποποιηθεί η γνωμοδότηση αυτή και αυτόν τον δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την οικολογική επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Στη δική μου χώρα ε, η αιωλική ενέργεια, ο κλάδος αυτός, ε, είναι δεύτερο σε απορρόφηση προϊόντων χάλιβα. Καταλαβαίνετε. Ε, επόμενος συνάδελφος, ο κύριος Παύρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο μήνυμα της κυρίας Φόρτ που δυστυχώς σχολείεται και αποσιάζει. Υποστηρίζω πλήρως τις ε, πρωτοβουλίες που κάνουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μείωση του γραφειοκρατικού άχθους και φόρτου στη βιομηχανία και στον κλάδο. Ιδιαίτερα ανησυχώ για τη διαφυγή ε, βιομηχανιών που παράγουν διοξίδιο του άνθρακα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε Επίσης και μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικές ε, τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν αρκούν οι δηλώσεις. Χρειάζεται και δράση με σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δράση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Λιωτάρ, παρακαλώ. Α, δεν θέλει να euh, Κυρία Λεπάζου, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι προαλήσαντες όπως ο Λάινεν, ο Γιου Λάινεν. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης στους τομείς εκείνους πραγματικά βρισκόμαστε η ηγετική θέση όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, για παράδειγμα, τα οποία βέβαια δεν καταφέραμε να μεταφράσουμε σε πραγματική βιομηχανική παραγωγή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στους τομείς αυτούς όπως οι πρώτε ύλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιμείνουμε σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνώ με τον προσανατολισμό της έκθεσης αυτής που νομίζω ότι στρέφεται περισσότερο στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Σίγουρα το ζήτημα της ενέργειας είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Δεν νομίζω πάντως ότι προωθώντας την προώθηση της ενέργειας η οποία έχει πάρα πολλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, ότι θα καταφέρουμε τελικά να επαναβιομηχανίσουμε την Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε τι νέε πηγέ ενέργεια και όλε αυτέ τι νέε τεχνολογίε που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και να δημιουργηθούν και τα εγώμενα φύ δίκτυα. Τώρα, πρέπει να σα πω ότι ε, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να επαναβιομηχανήσουμε την Ευρώπη. Η κυρία Κορτίνας Γκουτιέρας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας πω τα εξή. Δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο στη ζωή. Κατά την άποψή μου τώρα έτσι θα βλέπουμε, άσπρο-μαύρο. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πρώτον, η Ευρώπη έχει στόχους στο DNA της ήδη. Η αηφορία, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμιά αφεβολία επίσης ε, ότι το νερό θα πρέπει να είναι καθαρό, το περιβάλλον, να μειωθούν οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και μεταξύ άλλων για ένα λόγο. Η ίδια βιομηχανία θέλει να χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Είναι τεράστιο το κόστος στην Ευρώπη για την ενέργεια. Είναι και η πιο ακριβή ενέργεια. Ε, το 90%, το 90 της βιομηχανίας θέλει να εκπέμπει λιγότερο. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σφάλαμε, διότι οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα που έχουμε για τη μείωση ε, των εκπομπών δεν είναι εύκολο στην πράξη. Παράδειγμα, ε, έχουμε ποντάρει στην αφαλάτωση πριν από 10 χρόνια. Μαζικά, δυναμικά. Αλλά ποιος θα είχε φανταστεί τότε πόσο θα κόστιζε η ενέργεια. Είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα η αφαλάτωση που είναι στο κάτω-κάτω μία πρόταση οικολογική, καλή και χρήσιμη και ελπιδοφόρα για το μέλλον, δεν έχει βρει ακόμα τεχνολογία που να τρώει λιγότερη ενέργεια. Εάν καταφέρουμε, υπάρχουν απόπειρε προσπάθειες να ε, φτιάξουμε μονάδες αφαλάτωσης που να μην καταναλώνουν τόση ενέργεια, για να χρησιμοποιούμε και ανανεώσιμες, τότε μπορεί να συζητάμε για την αφαλάτωση. Σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει το κόστος ο καταναλωτής, ούτε εμείς να ε, επομιστούμε αυτό το τεράστιο κόστος που έχει και εκπομπές ε, μια μονάδα αφαλάτωσης σε λειτουργία. Τι εννοώ, να είμαστε λιγότερο γενικόλογοι και να μπαίνουμε σε κάθε τομέα, γιατί ο κάθε τομέας ε, χρειάζεται το χρόνο του για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν αμφισβητώ ε, ότι δεν πρέπει να, σκοτώσουμε τη βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι το μέλλον μας, αλλά ποια βιομηχανία και τι προϊόντα σε χαμηλό κόστος ε, παράγουν κάποιοι άλλοι με χαμηλούς μισθούς και με μεγάλη ρήπανση. Αυτό θέλουμε. Όχι. Θέλουμε βιομηχανία στην Ευρώπη. Δεν είμαι κατά της νομοδότησης. Χρειάζεται επεξεργασία. Η ιδέα δεν θα πρέπει να αλλάξει, αλλά οι χρόνοι να διαφέρουν για κάθε χώρα και για κάθε κλάδο και να ε, υποστηρίζουμε την καινοτομία γιατί πολλές χώρες δεν είναι σε θέση να το πράξουν αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. uh... Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι κάπως περίεργη. Όταν τη διαβάζω, μου δίνει την εντύπωση ότι ε, διαβάζω κάποιες, κάποια δόγματα της δεκαετίας του 50 και του 60 σοβιετικής φύσης. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται στο μέλλον της Ευρώπης. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε φτηνή ενέργεια, και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια χρηματοδότηση όσον αφορά την, ε, ιδιω... τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται, χωρίς όμως να υπάρχει επί τα πρόσβαση στις γνώσεις αυτές οι οποίες θα δημιουργηθούν. Ε, επίσης, ε, λέγεται ότι δεν θα, υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθεσία για τις κλιματικές αλλαγές η οποία να βάλει κατά τον ταγωνισμό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ατενίζουμε το μέλλον. Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία προωθούμε για το μέλλον θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την ενέργεια. Αυτό κάνουν και άλλες χώρες, Κίνα για παράδειγμα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ε, εμεί υιοθετήσουμε ουσιαστικά ένα παλαιό σοβιετικό σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταφέρνουμε απολύτω τίποτα δεν εστιάζεται στα σωστά σημεία η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να προωθήσουμε βιομηχανία στην Ευρώπη με την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να γραφτεί εξ αρχή η γνωμοδότηση αυτή και να δούμε πραγματικά ποιε περιβαλλοντικέ επενδύσει μπορούν να γίνουν στα πλαίσια τη επαναβιομηχάνηση Ευρώπη, που μπορούμε πραγματικά να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Εκεί έγκυται το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η όλη έκθεση θα πρέπει να εστιαστεί σε άλλα σημεία. Ο κύριο Χίπνερ το λόγο. Κύριε συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά τώρα με την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ευρώπη, θα πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες. Η καινοτομία, ναι, συμφωνώ. Οι νέες τεχνολογίες επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι σωστός στόχος. Το ερώτημα είναι όμως γιατί τα αποκαλούμε αυτά πράσινη οικονομία. Συμφωνώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί η πράσινη οικονομία, αλλά δεν είναι και η μοναδική οικονομία που διαθέτουμε. Πρέπει βέβαια να χρησιμοποιούμε με τρόπο βιώσιμο τους πόρους, αλλά να έχουμε και κάποια λογική. Πρέπει να αναπτύξουμε την καινοτομία και στα όσα έχουμε και με τους πόρους που διαθέτουμε. Στην Ινδία ή στην Κίνα, εκεί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους πόρους που διαθέτουν. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που ωστόσο είναι δύσκολο βέβαια να αναπτυχθεί εφόσον μετακινηθεί ολόκληρη η βιομηχανία μας και πάει κάπου στην Ασία. Πώς θα πείσουμε τους νέους μας να μείνουν εάν δεν δημιουργήσουμε συνθήκες διαβίωσης που να είναι ορθές. Εάν τελικά αγοράζοντας καταναλωτικά αγαθά που προέρχονται από αλλού, από το εξωτερικό, διώξουμε τελικά όλους τους νέους μας, ποιος θα μείνει εδώ δεν είναι μονάχα οι ανεμογεννήτριες. Ο χάλι μας χρειάζεται παντού. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσά δεν έχετε τεχνικό background. Αν αρνάζουμε τους νόμους κάθε τόσο, δεν θα βιώσει, δεν θα ζήσει η βιομηχανία μας, διότι κανένας δεν θα μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας, εφόσον αλλάζουμε διαρκώς τις συνθήκες. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως. Οφείλει να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη βιομηχανίας. Ορισμένοι μιλούν για μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Ναι, αλλά για ποιο λόγο, για ποιο σκοπό. Εμείς πρέπει επιτέλους να κάνουμε και έργα και όχι μόνο λόγια. Ως δημοκράτησα, δέχομαι, ε, σέβομαι μάλλον την άποψη του κ. Σιμάνσκι, αλλά ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος συμφωνώ με ορισμένους από τους συναδέλφους μου που είπαν ότι πρέπει να αποσύρουμε το κείμενο και να γράψουμε νέο. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε βέβαια με τροπολογίες έτσι ώστε να απηχεί τις απόψεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Γιατί η κυρία Χίπνερ έχω την εντύπωση ότι αυτό που ε, υποστηρίζει είναι ε, να συνεχίσουμε την βιομηχανική πολιτική του 19ου και του 20ου αιώνα. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτό. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στις προκλήσεις που μας τίθενται σήμερα. Δηλαδή, βεβαίως είναι θέμα να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησης στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους που αυτή τη στιγμή βασίζονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αλλά όχι με την έννοια ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτές, αλλά να καταστήσουμε δυνατόν στις βιομηχανίες αυτές να προσαρμοστούν σε εναλλακτικέ επιλογές. Και όχι αυτές που ε, ε, αναφέρονται εδώ ως φθηνές, διότι μίλησε η κυρία, ε, ο κύριος Σιμάσκη για το «fraking», αλλά αυτά όμως είναι μορφές ενέργειας της, του παρελθόντος. Εδώ χρειάζεται λοιπόν έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτό το fracking, δηλαδή η ε, εκμετάλλευση του πετρελαίου που βγαίνει από το σχιστόλιθο, πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Εφόσον δεν μιλούμε και για την πυρηνική ενέργεια, πρέπει να δούμε το κόστος της ενέργειας αυτής αναμονάδα μέχρι και την ανακύκλωση των καταλήπων. Εγώ αναμένω τις τροπολογίες διότι όπως είναι το έγγραφο δεν μπορεί να απηχεί την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πολλοί συνάδελφοι δήλωσαν ότι θα ε, τίνουν χείρα βοηθείας δια των τροπολογιών για τη βελτίωση της εκθέσεως του κ. Σιμάνσκι. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά της βαρύτερης οικονομικής κρίσης της μεταπολεμικής περίοδου. Πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πραγματικά πώς θα προχωρήσουμε. Η πράσινη οικονομία νομίζω ως ορολογία τελικά θα καταργηθεί, διότι κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει τι μπορεί να σημαίνει. Και στους Ρίο πάλι δεν συμφώνησαν. Ολόκληρη η οικονομία πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί με τρόπο βιώσιμο και όχι μόνο οικολογικά αλλά και οικονομικά διότι η οικονομική κρίση προκύπτει από μια βαρύτατη δημοσιονομική κρίση. Πρέπει και για αυτό να αγωνιστούμε αλλά και για την επί το ανθρωπινότερο διαμόρφωση των συνθήκων εργασίας, τις κοινωνικές συνθήκες δηλαδή αυτό ο χωρισμό σε δίθεν πράσινη οικονομία και δήθεν καφετιά οικονομία δηλαδή των ορεικτών καυσίμων δεν μπορεί να είναι σωστός. Χάλιβα, χημεία κλπ. Όλα πρέπει να λάβουν με τον τρόπο αυτό. Γιατί είναι τόσο πετυχημένη η μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης λόγω δίθεν της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος. Όχι. Πληρώνουμε στη Γερμανία τη δεύτερη υψηλότερη ανά τον κόσμο τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι άλλοι λόγοι. Λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τον κύριο Σιμάνσκι να διορθώσει την έκθεσή του. Βλέπω ότι ο κύριο Σιμάνσκι χαμογελά και νομίζω ότι όλοι θα βοηθήσουν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο θα λάβει το λόγο. Καλά. κανείς. Έχουμε κάποιον κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, εμείς συντάξαμε την ανακοίνωση αυτή μετά από την κρίση και γι' αυτό έχουμε βασιστεί σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες. Πρόσβαση ε, σε χρηματοδότηση, δεξιότητες, καινοτομία και ε, διεθνές εμπόριο. Είδαμε ότι η λίγη ανάπτυξη που έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα προέρχεται από τις εξαγωγές, δηλαδή από ανάπτυξη η οποία συμβαίνει στην ουσία εκτός Ευρώπης. Να έλθω σε αυτό που είπατε για την καινοτομία, που είναι και η βασική γραμμή της ανακοίνωσης και όχι μόνο έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και η χρήση πραγματικά αυτής της ε, καινοτομίας. Και γι' αυτό έχουμε βάλει έξι προτεραιότητες από τις οποίες και οι έξι στοχεύουν σε αυτό το πρασίνισμα της βιομηχανίας που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καθαρότερα αυτοκίνητα, προϊόντα βασισμένα σε μια βιολογική παραγωγή και νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε ιδιαίτερα και στις βασικές συνθήκες πλαίσια, όχι μόνο το πρασίνισμα, όπως είπαν και οι περισσότεροι από εσά εδώ, βλέπουμε και εμείς το πρασίνισμα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ευχαριστώ εσείς τώρα κύριε Σιμάνσκι, γιατί ο Επίτροπος αναμένει πρώτων πυλών. Θέλετε να απαντήσετε ή... Ναι, θέλω πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και ευχαριστήσεις προς όλους τους ε, προλαλήσαντες. Είχα επίγνωση του γεγονότος ότι θα κατατεθούν κάποιες ε, τροπολογίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει να σφυριλατήσουμε ένα συμβασμό. Ε, ούτε αυτό που λέει κανείς σε μια γνωμοδότηση είναι απόλυτο, έτσι, χαραγμένο στο μάρμαρο. Και καμιά φορά μπορεί κανείς να ε, παραδέχεται ότι ε, χάνει. Ε, ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ την Πολωνία και έχουμε άλλη αντίληψη και άλλη εικόνα, ίσως διαφορετική από τη δική σας για τη βαριά βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήθηκε εδώ η μερίσια διάταξη. Είπαμε προθεσμία 15 του μηνός, 19 Ιουνίου θα ψηφίσουμε εδώ και 26 Σεπτεμβρίου στην Ήτρε και στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα ψηφιστεί. Και πάμε στο επόμενο θέμα τώρα και καλωσορίζουμε τον ε, κύριο Αντώνιο Μπορ στην Ομίγυρη, Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Υγείας. So, jetzt können wir starten. Αρχίζουμε. Καλωσορίζω και πάλι θερμότατα ε, τον Επίτροπο ε, Αρμόδιο για θέματα δημόσιας υγείας. Ε, θα του δώσω το λόγο για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα μπούμε στη συζήτηση. Πρώτα θα μιλήσουν οι συντονιστές και μετά όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν ερωτήσεις όσοι θέλουν. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη που μας απασχολούν και πρέπει να επεξεργαστούμε. Κοιτάω την κυρία Λίντα Μακέβεν, έχουμε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού που αποτελεί για μας μεγάλο φόρτο εργασίας. θέλουμε να ευοδοθεί και χαιρόμαστε ε, που ε, τέλειωσε αυτό πριν τα Χριστούγεννα με όλα τα δεινά της αλλαγής χαρτοφυλακίου κτλ. Ε, μετά έχουμε την έκθεση Λίζε και Ντάγμα Ροτ Parent για την in vitro διαγνωστική και ιατροτεχνικά βοηθήματα. Έγιναν και διάφορα σεμινάρια, εργαστήρια. Είναι μεγάλη η υπόθεση αυτή που πρέπει να ρυθμιστεί και που μας απασχολεί πάλι. Και έχουμε και την έκθεση κυρίας Γκλένης Βίλμοντ για τις κλινικές δοκιμές. πάλι και αυτό είναι ένα θέμα. Ο Ζιλ Παρνιό, να πω και κάτι ευχάριστο, μας ανακοινώνει ότι υπήρξε μια θετική εξέλιξη, μια συμφωνία για ε, τη διασυνοριακή συνεργασία για θέματα ασθενών. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που έχουμε στη μερική διάταξη, αλλά περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει και νέες προτάσεις ε, για να προετοιμαστεί η νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Βέβαια δεν θα προλάβουμε εμείς να τα ε, επεξεργαστούμε. Ένα ε, νέο κανονισμό τελών για την αίμα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Θέλουμε να συγχρηματοδοτούνται οι οργανισμοί και όχι σε εξαετή, επταετή ε, προγράμματα να είναι χρηματοδότηση, να είναι αυτοτελείς, ανεξάρτητοι οι οργανισμοί αυτοί και αυτό σημαίνει κατά την άποψή μου και αυτοχρηματοδοτούμενοι κατά κάποιο τρόπο ε, λογικό για να μπορούν να καλύπτουν και τα όσα τους έχουμε αναθέσει. Αυτό δεν αφορά μόνο τον οργανισμό φαρμάκων αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θα είναι πιο, πολύ σημαντικό. Αυτά και σταματώ εδώ. Δεν θέλω να βγάλω λόγο. Να δώσω το λόγο μέσα στον Επίτροπο. Παρακαλώ κύριε Πώς. Thank you, Mr. Chairman. This is, I my... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Πράγμα το οποίο καταδεικνύει πόσα πολλά ζητήματα τελικά καλύπτονται από τη δική σας την Επιτροπή και από τις δικές μου τις ε, αρμοδιότητες. Όντως είχαμε τις ακροάσεις στις οποίες αναφερθήκατε και έχουμε έπειτα και τον διάλογο αυτό τον διαρθρωμένο με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο οποίος παρακολουθεί κάθε φορά τις εξελίξεις που έχουμε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Ξέρετε βέβαια ότι η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται το Μάιο του 2014, επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτή είναι ευχή τόσο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιταχύνουμε κάπως τι εργασίε μα κατά τη διάρκεια του τρέχοντο έτου και χαίρομαι πάρα πολύ με τον τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει την οδηγία για τα καπνά, για τα πρώτα καπνού. Και βέβαια αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει επισκιάσει άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία. Θεωρώ ωστόσο ότι το, η υγεία αυτή είναι ιδιαίτερα καλά ισοσκελισμένη, ισορροπημένη. Σίγουρα κάπου μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό όμω να καταφέρουμε να εγκρίνουμε κατά τη διάρκεια τη τρέχουσα νομοθετική θητεία. Και δεν σας λέω, δεν αποκαλύπτω κάποιο μυστικό όταν σας λέω ότι αυτοί οι οποίοι αντιτάσσονται στην οδηγία αυτή δεν αντιτάσσονται ευθέω στην οδηγία, λέγοντας ότι δεν δέχονται κάποια σημεία της, αλλά ότι προσπαθούν ουσιαστικά να επιβραδύνουν τη διαδικασία έγκρισής της. Όσοι όμως είμαστε υπέρ της ισορροπημένης αυτής προσέγγισης για μεγαλύτερη ρύθμιση των προϊόντων καπνού, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα αυτή, μπλοκαρίσματο δηλαδή τη οδηγία και θα πρέπει εμεί να αντιταχθούμε σε κάτι τέτοιο. Και όταν συζητούσαν πριν μερικέ εβδομάδε ε, την έκθεση τη κυρία Μακέβεν, ε, ακούστηκαν πολλέ διαφορετικέ απόψει και ορισμένοι μάλιστα θέλαν ακόμα και πιο αυστηρά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπονται αυτή τη στιγμή. Και ότι θα πρέπει να καλύπτονται και κάποια νέα καινοτόμα προϊόντα στα πλαίσια των προϊόντων καπνού και θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια οδηγία η οποία θα έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογή και θα καλύπτει πάρα πολλέ πτυχέ των πρώτων καπνού. Προσβλέπω πάντως πολύ θετικά στα αποτελέσματα των δικών σας των συζητήσεων που πραγματικά θα συμβάλλουν πάρα πολύ στη σημαντική αυτή οδηγία η οποία πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις επόμενες γενναίες. Θεωρώ ότι μέσω της οδηγίας αυτής ο αριθμός των καπνιζόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί κατά 2% σε περίοδο, σε περίοδο 5 ετών. Δηλαδή 2 εκατομμύρια λιγότεροι καπνιστές, πράγμα το οποίο σημαίνει καλύτερη υγεία για τους πολιτές μας, αλλά και εξοικονόμηση επίσης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις κυβερνήσεις μας όσον αφορά τις θεραπείες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις παθήσεις που προκύπτουν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και όλους ιδιαίτερως την εισηγήτρια για τις παρατηρήσεις της και ελπίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε μια φιλόδοξη οδηγία για τα πρώτα καπνού πολύ σύντομα. Τώρα όσον αφορά το κρέας αλόγου. Ας περάσουμε στο επεισόδιο τώρα αυτό. Τι συνέβη από την τελευταία φορά που σας μίλησα. Νομίζω ότι ήταν το Φεβρουάριο η τελευταία φορά που σας είδα στην Επιτροπή σας. Σας είχα υποσχεθεί τότε ότι μόλις είχαμε τα αποτελέσματα από τις δοκιμές DNA που γίνονται τόσο για την παρουσία λογίσιου κρέατος στο βόλιο κρέας, όσο επίσης και τη χρησιμοποίηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στο κρέας αλόγου, ότι θα δημοσιεύαμε, θα κοινοποιούσαμε αμέσως τα αποτελέσματα. Και το είπα αυτό προτού να γνωρίζω τελικά τα αποτελέσματα, γιατί νομίζω ότι μόνο μέσω της διαφάνειας θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στα νομοθετήματά μας. Και ακριβώς λοιπόν αυτό έπραξα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε τις μελέτες οι οποίες γίνανε και μολονότι πρόκειται απλώς για συστάσεις που κάνουμε στα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη ακολούθησαν τις συστάσεις αυτές και κάνανε και περισσότερα πράγματα, όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Ενώ ε, προβλεπόταν να γίνουν απλώς 250 δοκιμές, γίνανε πολύ περισσότερες. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, εξέτασαν όλα τα σφαγεία αλόγων σφάγε, με συγχωρείτε, λόγων, ακριβώς για να δούνε αν τελικά υπήρχαν φάρμακα στο κρέας τους. Και νομίζω ότι πολλά άλλα κράτη-μέλη κάναν το ίδιο πράγμα. Και δημοσιεύθηκαν όλα αυτά τα αποτελέσματα μέσα σε 24 ώρες. Η καταληκτική προθεσμή ήταν η 15η και στις 16 του μηνός είχαν δημοσιευθεί όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και ξέρετε ότι από τις δοκιμές ε, επιβεβαιώθηκε πραγματικά το ότι δεν επρόκειτο για ένα θέμα δημόσιας υγείας και τρία μόνο κράτη-μέλη είδαν ότι υπήρχαν συγκεκριμένα φάρμακα στο αλογίσιο κρέας, δηλαδή λιγότερο από 0,5% του συνόλου των δειγμάτων που εξετάστηκαν. Τώρα όσον αφορά την ε, παρουσία αλογίσιου κρέατος με λανθασμένη σήμανση ουσιαστικά, τα ποσοστά ήταν κάτω του 5%. Βέβαια το 5% μπορεί να θεωρηθεί ε, σημαντικό ποσοστό παρόλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά το ποσοστό ήταν περιορισμένο στο 5% ή κάτω του 5%. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, ο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών λειτουργήσε πολύ καλά. Τα κράτη-μέλη κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ε, τι απατηλέ αυτέ επιχειρηματικέ διαδικασίε που είχαν εντοπιστεί σε ορισμένε περιπτώσει. Τώρα, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα στο μέλλον. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, τι διδάγματα έχουμε αποκομίσει υπό το φως της εμπειρίας αυτής. Όπως λέγεται και στο σχέδιο δράσης το οποίο σας απέστειλα κύριε Πρόεδρε στι 20 ε, Μαρτίου θα επικεντρωθούμε σε τρία σημεία. Πρώτον, να ενδυναμώσουμε τις ικανότητές μας προκειμένου να καταπολεμήσουμε την απάτη στο τομέα των τροφίμων, να έχουμε επίσης πιο ε, έντονου ελέγχου και κυρώσει. και τρίτον, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε όσον αφορά τα λεγόμενα διαβατήρια για το αλογίσιο κρέα. Ξέρετε ότι ε, Ήδη έχουν ξεκινήσει, μάλλον έχουμε δημοσιοποιήσει μια επίσημη δέσμη μέτρων για τον έλεγχο του αργοδιατροφικού τομέα. Χθε μάλιστα κινητοποιήθηκε, ε, δημοσιοποιήθηκε με συγχωρείτε, η δέσμη αυτή και στα πλαίσια των νομοθετημάτων αυτών προβλέπεται ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για την απατηλή αυτή δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα κυρώσεις οι οποίες ουσιαστικά θομοιάζουν με τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα κάθε φορά που εντοπίζονται φαινόμενα απάτης. Όλα λοιπόν αυτά τα φαινόμενα απατηλής σήμανσης ουσιαστικά θα επιφέρουν πλέον πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Ας περάσουμε τώρα στις τέσσερις ε, τομεακές ε, προτάσεις που θα απλουστεύσουν και θα δυναμώσουν τελικά την νομοθεσία την οποία έχουμε στην ε, αγροετροφική αλυσίδα. Χθε δημοσιοποιήθηκε η πρόταση αυτή και είπαμε ότι αντί να έχουμε 70 διαφορετικές ρυθμίσεις εθνικές όσον αφορά τον αγροετροφικό τομέα θα έχουμε 5 μόνο και χθε εγκρίναμε και μία δέσμη μέτρων η οποία προβλέπει μία προσέγγιση η οποία θα βασίζεται περισσότερο στην ανάλυση του κινδύνου όσον αφορά την προστασία της υγείας των τροφίμων και των ζώων και μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα πλαίσια της αγροτροφικής αλυσίδας. Θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποια εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε περισσότερο στους κινδύνους που εμφανίζονται στα πλαίσια του αγροτροφικού τομέα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο όλης της αγροτροφικής αλυσίδας αλλά ακόμα και των εισαγόμενων προϊόντων. Να πω κάποια πράγματα τώρα και για τους ίδιους τους σπόρους, γιατί και για αυτούς μιλάμε τελευταία. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες ε, φήμες και απεστάλησαν μάλιστα και κάποιες επιστολές, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενδυναμώσει τον τομέα των ε, σπόρων, της βιομηχανίας των σπόρων και ζητά μάλλον ότι προσπαθεί να επιβαρύνει τον τομέα αυτόν, ζητώντας περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και το καθεξής. Αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά άδικο και προφανώς ασφαλμένο. Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, όλοι οι σπόροι πρέπει να καταγράφονται. Μετά τη νέα όμως αυτή νομοθεσία και την έγκρισή της, οι παραδοσιακοί σπόροι θα έχουν ένα πιο ελαφρύ καθεστώς καταγραφής. Για παράδειγμα, δεν θα απαιτείται κάποια δοκιμή ή κάποιο τεστ προκειμένου να καταγραφούν αυτοί οι παραδοσιακοί σπόροι. Και όσον αφορά τους νέους σπόρους που έχουν να κάνουν με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για αυτούς δεν θα προβλέπεται καμία υποχρέωση καταγραφής, ενώ τώρα δεν γίνεται καμία διάκριση στην υφιστάμενη νομοθεσία ανάμεσα στους παραδοσιακούς και τους νέους σπόρους. Επομένως, και αυτοί οι νέοι σπόροι των μικρών επιχειρήσεων πρέπει να καταγράφονται, υπόκεινται στο ίδιο καθεστώ. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε την ε, κατηγορία αυτή ότι ε, επιβαρύνουμε περισσότερο με γραφειοκρατικές διαδικασίες τον τομέα των ε, σπόρων. Τώρα, όσον αφορά τα τέλη καταγραφής για τη βιομηχανία των σπόρων. Με τη νέα νομοθεσία προβλέπεται ότι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα εξαιρούνται πλήρως από οποιοδήποτε τέλος για οποιοδήποτε σπόρο. Επομένως δεν θα προβλέπονται καθόλου τέλη για οποιαδήποτε καταγραφή σπόρων αν η αίτηση έχει υποβληθεί από μία πολύ μικρή επιχείρηση. Ακόμα και για τους παραδοσιακούς σπόρους θα προβλέπετε ότι τα τέλη καταγραφής, καταχώρησης θα είναι πολύ μικρότερα από αυτά που τα οποία ισχύουν τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί να συμφωνεί κανείς με τη νέα αυτή νομοθεσία, μπορεί κάποιος να αντιτάσσεται στη νομοθεσία αυτή, αλλά τα πράγματα έχουν ε, έτσι ουσιαστικά δεν είναι διαφορετικά. Και στη νέα αυτή νομοθετική δέσμη προβλέπονται οι νέες αυτές διατάξεις. Έτσι θα έχουν τα πράγματα στο μέλλον και δεν θα ισχύουν οι πρώτερες νομοθετικές διατάξεις που είχαμε στο παρελθόν. Ήθελα να στείλω το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα ότι για τους παραδοσιακούς και τους νέους πόρους έχουμε μια νέα νομοθεσία με λιγότερες υποχρεώσεις καταγραφής, με χαμηλότερο κόστος που ουσιαστικά ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος που βαρύνει τις επιχειρήσεις. Τώρα όσον αφορά τα νέα τρόφιμα και την κλωνοποίηση. Όσον αφορά τις ε, επόμενες προτάσεις, θα γνωρίζει και η κυρία Λιωτάρα αλλά και άλλοι οι ότι πραγματικά δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποια συνένεση στα πλαίσια της ε, συνεδρίασης που έγινε το Μάρτιο 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως είχε την πρόθεση να προτείνει μια νομοθεσία για τα κοινοτρώμα τόφημα, καθώς επίσης και την κλωνοποίηση των ε, ζώων. Όσον αφορά το τελευταίο αυτό ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ευρεία διαβούλευση προσπαθεί ουσιαστικά να ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή μία μελέτη αντικτύπου και θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε επίσημη πρόταση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή αξιολόγηση αντικτύπου. Όσον αφορά τα καινοτόμα τρόφιμα, υπάρχει μια Γενική Συμφωνία του Μαρτίου 2011. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Όσον αφορά του γενετικά τροπημένου οργανισμού, θέλουμε να σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά την πρόταση καλλιέργεια. Ξέρετε ότι η κυρία Λαπάζη είναι η αρμόδια εισηγήτρια. Πρόταση η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο. Έχω ήδη προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με τα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αντιδράσεις που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη, κάποιους ενδιασμούς που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο το μοθετικό αυτό Θέλω πραγματικά να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο, να ξεπεράσουμε το εφιστάμενο αδιέξοδο και πιστεύω ότι μέσω της νέας αυτής πρότασης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς τα κράτη-μέλη θα μπορούν πλέον ελεύθερα να επιλέγουν αν θέλουν ή όχι να καλλιεργούν στην επικράτειά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και για άλλους λόγους, όχι μόνο περιβαλλοντικούς. Όσον αφορά τώρα τις ιατρικές συσκευές, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο νέος επίτροπος από την 1η Ιουλίου θα αναλάβει το ζήτημα αυτό. Βέβαια, στο διάμεσο διάστημα εγώ ασχολούμαι ακόμα καθότι βρίσκεται στα πλαίσια των δικών μου αρμοδιοτήτων. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουμε στον τομέα αυτό και βέβαια να εξασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη αλλά και την υγεία και την προστασία του κοινού, ιδίω υπό το φως κάποιων πρόσφατων σκανδάλων. Θέλουμε να ενισχυθούν περισσότερο οι κανόνες όσον αφορά την παρακολούθηση από την αγορά, όσον αφορά την παρακολούθηση ακολούθησε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα μέτρα αυτά όμως θα πρέπει να είναι αναλογικά προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει πραγματικά στην πρώτη γραμμή της καινοτομία των ιατρικών συσκευών, ένα τομέα ο οποίο τελικά δημιουργεί και περισσότερε θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω θα γνωρίζετε, δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή ένα σύστημα πρώτερης φαρμακευτικής έγκρισης για τις ιατρικές αυτές συσκευέ, γιατί θεωρούμε ότι θα δημιουργούσαμε μεγαλύτερο κόστος και διοικητικό άκθος και ότι δεν θα προωθούσαμε καθόλου τον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό εξέτασης και ελέγχου προκειμένου να μπορούν να ενημερώνουν οι αρμόδιες αρχές και να υποβάλουν κάποια γνωμοδότηση προτού μία ιατρική συσκευή ψηλού κινδύνου τεθεί στην αγορά αλλά και αφού τεθεί στην αγορά. Ο τομέας αυτός αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα για μένα και πραγματικά θα ήθελα να πετύχουμε μία συμφωνία πολύ σύντομα στον τομέα αυτό. Όσον αφορά τώρα τις κλανικές δοκιμές, ως προς αυτό χαίρομαι για την πρώτη αντίδραση που υπήρχε στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ όμως σε τέσσερα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει κάποια ανησυχία. Όσον αφορά τις δεοντολογικές επιτροπές και την γενικότερη δεοντολογία, η πρόταση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να, εξεράσει, να εξαιρέσει με συγχωρείτε, τις επιτροπές δεοντολογίας από τις κλινικές δοκιμές που θα γίνονται. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να παρακάμψω τον τομέα της δεοντολογίας από την πρόταση αυτή. Δεν θα θέλαμε πάντως η πρόταση αυτή να είναι γνωστή μόνο για την πτυχή της αυτή που θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο. Επομένω μπορούμε να δεχθούμε οποιαδήποτε πρόταση ενισχύει την δεντολογική διάσταση της πρότασης, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πρόκειται για κανονισμό και όχι οδηγία. Επομένως δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τη λειτουργία μιας Επιτροπής Δεντολογίας. Επίσης θα πρέπει να είναι εντελώ ενσωματωμένη διαδικασία διοντολογική στην κύρια διαδικασία και να μην αποτελεί μια ξεχωριστή παράλληλη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα την διαφάνεια των κλινικών δοκιμών, πάλι εδώ πέρα θα προβλέπετε ότι μετά, μια, μετά την δοκιμή θα υπάρχει μια πλήρης μελέτη η οποία θα, θα δημοσιοποιείται. Όσον αφορά τι κλινικέ δοκιμέ τώρα στι τρίτε χώρε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τη δική, δική μα νομοθεσία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι οι κλινικές αυτές δοκιμές θα γίνονται ακολουθώντας τους γενικότερους κανόνες που ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τα προτινόμενα κριτήρια για του συμμετέχοντες κλινικέ δοκιμέ. Προβλέπονται εδώ πέρα κριτήρια για την προστασία των ασθενών και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύουν πάλι κάποιοι κοινοί κανόνες. Θα πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εφιστάμενη εργασία για την οδηγία των κλινικών αυτών δοκιμών κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης νομοθετικής θητείας. Όσον αφορά τώρα τους τις διασυνοριακές απειλές στην υγεία, Χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια συμφωνία για την νομοθεσία αυτή, η οποία θα προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες από, μια μεγάλη, από ένα μεγάλο αριθμό διασυνοριακών απειλών στην υγεία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα κράτη-μέλη δέχονται σε θελούσια βάση να συμμετέχουν σε μια κοινή διαδικασία δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τα εμβόλια. Και σε μια θελούσια βάση θα υπογραφεί μια συμφωνία ε, κατά τη διάρκεια της πληθωνικής προεδρίας. Κατά αυτόν τον τρόπο όλες οι χώρες θα μπορούν να έχουν ασφαλή εμβόλια. Τώρα, πρόγραμμα για την υγεία. Πρωτού ολοκληρώσω, θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ και στο πρόγραμμα για την υγεία, για το οποίο θα αρχίσουν πάλι οι συζητήσεις αφού ληφθεί κάποια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βασίζομαι πάρα πολύ στην δική σας Επιτροπή και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε μέχρι τα τέλη του έτου σε μια συμφωνία για το πρόγραμμα αυτό υγείας. Τώρα, όσον αφορά για τη γενική παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, ξέρετε ότι η οικονομική κρίση έχει, δημιουργήσει, έχει οδηγήσει σε περικοπές στον τομέα της υγείας σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Και όπως είπα στους υπουργού Υγείας, μην περιμένετε οι περικοπές αυτές ε, στον προπολογισμό στα κράτη-μέλη να μην επηρεάσουν τελικά και τους προπολογισμούς υγείας. Έχουν επηρεάσει και τον ίδιο τον προπολογισμό της ε, αρμόδιας διεύθυνσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας αρρωγής εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Προσπαθούν τα προγράμματα αυτά να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις που έχουν πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διάφορες χώρες και θέλουν ουσιαστικά να δημιουργήσουν μια πιο ορθολογική χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών. Και πολλέ βέβαια από τι μεταρρυθμίσει αυτέ έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη προτού εμφανιστεί η οικονομική κρίση. Τα μέτρα λοιπόν έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, καθώς επίσης και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η DG ECFIN βρίσκεται στην πρώτη θέση της διαδικασίας αυτής, ενώ οι δικές μου υπηρεσίες συμμετέχουν σε αποστολές της Τρόικας κάθε φορά που συζητάνε ζητήματα δημόσιας υγείας και ε, ε, προσφέρουν ε, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη κάθε φορά που ζητάτε κάτι τέτοιο. Και βέβαια εμείς σεβόμαστε απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να δυναμώσουμε τα συστήματα υγείας των κρατών μελών και να καταφέρουμε τελικά να επικεντρωθούμε στις βασικές αξίες και αρχές που πρέπει να έχουμε σε ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Καθολικότητα, ισότητα και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Για παράδειγμα, στο μνημόνιο κατανόησης για την Κύπρο είχαμε πει ότι η Κύπρος θα πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο επίπεδο προκειμένου να υπάρχει μια μελλοντική επέκταση αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εξαρτάται τελικά από την υγειονομική ιδιωτική παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κάλεψα πολύ γρήγορα κάποια σημαντικά ζητήματα που είναι επιτάπητος αυτή τη στιγμή. Προσβλέπω στις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ πολύ για την πλήρη εικόνα που δώσατε για όσα θέματα ε, εκκρεμούν και όσα θέματα ε, πρόκειται να συζητηθούν ακόμα και ιδίως για το υλικό σπόρων που η στη χώρα μου έχει ήδη γίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν θέλει να απαγορεύσει τη χρήση κάποιων σπόρων. Εγώ μίλησα με δημοσιογράφους. Ξεκίνησε μια είδηση στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα και αυτό που έκανε οι δημοσιογράφοι είναι ότι την αντέγραψαν. Εγώ το βρίσκω απίστευτο ότι ορισμένα πράγματα δεν τα ελέγχουν πλέον, δεν τα διασταυρώνουν, απλώς τα αντιγράφουν. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ που είπατε για το θέμα αυτό ξεκάθαρα λόγια. Και αυτό και χαίρομαι που συζητούμε με την Κομισιόν πριν να υποκύψουμε στα μηνύματα αυτά των σιρήνων που ε, μεταδίδουν μηνύματα τα οποία δεν ή διαδίδουν μηνύματα τα οποία δεν έχουν διασταυρώσει. Τώρα θα προσπαθήσουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Πρώτα θα μιλήσει Ορισμένοι συνάδελφοι θα κάνουμε μια διάλειμμα, ένα διάλειμμα, θα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Frau Roth-Behrendt, Corinne Lepage, Esther de Lange, äh, Michel Rivasi, Jana Koudakis, Taylor, Pagnot, Okoni, Lier, äh, ε, Mas, äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, Äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? ξέχασα κανένα όνομα. Όχι, εντάξει, τότε λοιπόν είπα το όνομά σας. Την κυρία Γιάννα Κουδάκη. Δεν θα τολμούσα ποτέ να μην σας δώσω το λόγο. Έστω και αν... Έστω και αν εμφανιστήκατε σήμερα με άλλο φλιτζάνι στην Επιτροπή. Τώρα, για δύο λεπτά οι συντονιστές μετά θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος. Κύριε Πέτερ Λίζε πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε για την θετική συνεργασία από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας και ευχαριστώ επίσης για την έγκαιρη υποβολή της προτάσεως για τα προϊόντα καπνού που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα είναι σοβαρή η συζήτηση, ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και τροπολογίες ώστε να προχωρήσουμε και με την συναπόφαση και με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια πριν από τις ε, διακοπές. Επίσης για την κλωνοποίηση χαίρομαι που θα μας υποβάλλετε εγκαίρως πρόταση και να κάνετε την απαραίτητη πίεση στην Κομισιόν, να ασκήσετε στους άλλους ε, δηλαδή, επιτρόπους. Τώρα για τις εργασίες της Κομισιόν στην Τρόικα των χωρών που ε, πλήττονται από τη δημοσιονομική κρίση. Στην, στο έντυπο Lancet διαπιστώνουν οι συντάκτες της μελέτης ότι στις χώρες αυτές που πλήττονται από τη δημοσιονομική κρίση σημειώνονται αυξήσεις των ασθενειών, των νόσων και των αυτοκτονιών, ιδίως Πορτογαλία και Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγεται στο, στην μελέτη αυτή, στο άρθρο, αυτό, ότι η Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, δεν έχει λάβει υπόψη τη τα αποτελέσματα αυτά τη πολιτική που ασκεί. Ίσως πρέπει να τα διατυπώσουμε τα πράγματα αυτά με μεγαλύτερη ακρίβεια και σας παρακαλώ να δείξετε και θάρρος και απέναντι στους διαπραγματευτές της Τρόικα να ληφθεί υπόψη περισσότερη τεχνογνωσία που προκύπτει από την πολιτική υγείας. Είναι πραγματικά παράξενο ότι τον Ιανουάριο φέτος αποφασίστηκε για πρώτη φορά οι εφοπλιστές να πληρώνουν φόρους. Ταυτόχρονα γίνονται περικοπές στα συστήματα υγείας ήδη από την αρχή των παρεμβάσεων της Τρόικα. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να γίνουν καλύτερες περικοπές, καλύτερες εξοικονομήσεις. Ακούω για παράδειγμα ότι στην Ελλάδα υπάρχει διπλάσιος αριθμός γιατρών από το μέσο όρο των χωρών του ΩΣΑ. Μέχρι πού θα πάνε αυτές οι ε, διευκολύνσεις ή αυτές οι περικοπές η, η κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε για τον καπνό. Και εμείς δουλεύουμε σκληρά ε, και εγώ και οι Σάντο και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου για να προλάβουμε να ψηφίσουμε πριν από τι θερινέ διακοπέ και επομένω να προχωρήσει το θέμα και πριν από τη λήξη τη θητεία του παρόντο Κοινοβουλίου. Και για τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα το ίδιο. Έχουμε αύριο την λήξη τη προθεσμία τη καταθέσεω τροπολογιών. Τα πράγματα λοιπόν πηγαίνουν όπω προβλέπονται. Για να σε ερωτήσω τώρα για την υγιεινή των κρεάτων. Μιλήσατε για το πακέτο μέτρων για την υγεία των φυτών, αλλά για το κρέας Ακούω τώρα ότι η σχετική σας ανακοίνωση καθυστερεί και θα πάει πεντατέλη του έτους. Γιατί? Εδώ χρειάζεται κάποια προσοχή, διότι μιλείτε τώρα για νέα κατανομή χρονική των ελεγχών κτλ. Αυτό που ακούω όμως από τους επιθεωρητές είναι ότι από το 2006 τα ε, εργοστάσια που κόβουν το κρέας και το πακετάρουν είχαν επιθεωρήσεις κάθε μέρα. Αυτό άλλαξε. Άλλαξε μετά από την μεταρρύθμιση του 2006 και οι επιθεωρήσεις γίνονται τώρα. Ξέρω ότι θα αλλάξετε αυτό με τους προαναγγελθέντες ελέγχους. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να το σκεφτείτε πολύ προσεκτικά, διότι όλη αυτή η δεοντολογία για την τελευταία δεκαετία της Επιτροπής είναι μείωση των επιθεωρήσεων, μεγαλύτερη ανάλυση ευθύνη από τις εταιρείε. Αυτό όμως δεν είναι καλό. Δεν αρκεί να γίνονται επιθεωρήσεις τακτικά, έλεγε τακτικά για τρει μήνες όταν σημειώσετε ένα σκάνδαλο. Τι γίνεται όταν περάσει ο πανικός. Χρειαζόμαστε ένα καθεστώς το οποίο να είναι στέρεο και για μακρά διάρκεια. Εγώ φοβούμαι ότι καθυστερεί το πακέτο διότι αναμένουν όλοι να κατασυγάσει ο θόρυβος. Έτσι όμως χάνουμε από τα μάτια μας τους στόχους και θα παρακολουθήσουμε πάντως εμείς πάρα πολύ προσεκτικά το τι θα προτείνουν οι υπηρεσίες σας. Chris Evans. Chris Davis. Chris Δύο πράγματα για τις μέλησες πρώτα και για το τον περιορισμό της χρήσης νέο νοικοτινοειδών, νέο νίξ τα λένε αυτά, σε ε, για τις μέλισσες και το καλωσορίζω. Πραγματικά είναι η αρχή της προφύλαξης σωστά εφαρμοσμένη. Αλλά αυτοί ε, οι περιορισμοί είναι διετής. Και πώς θα το μετρήσετε μετά επιστημονικά για να αποδείξετε αν έχει αποδώσει το μέτρο ή όχι. Μέσα σε μια διετία. Αν ευθύνονται πραγματικά τα νέο ε, νικοτινοειδή για τη μείωση του αριθμού των μελισσών. Ε, και θα χρησιμοποιηθούν κάποια άλλα σκευάσματα συνθετικά ε, παραθροειδή, Πυρεθροειδή. Ε, χρειάζεται όμως κάποια επιστημονική απόδειξη όλο αυτό το θέμα. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο δύσκολο αυτό να αποδεχτεί μέσα σε μία διετία, όταν αυτή εκπνεύσει τι θα γίνει. Ε, υποθέτω ότι θα ζητήσετε ε, παράταση των περιορισμών αυτών μετά. Και πολύ σύντομα για τα καλλιντικά. Τώρα έχουμε μια συνολική απαγόρευση για την απαγόρευση πειραμάτων σε ζώα Ωραία. Πώς θα επιβάλλετε όμως ε, την ε, τήρηση ε, αυτών και στις εισαγωγές και στις κοινοτικές παραγωγές. Ο, ο κύριος Σλούτερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αν σας κατάλαβα σωστά, για τα προϊόντα καπνού τι είπατε. Αν προχωρήσουμε στο νέο πακέτο λοιπά. Ε, δεν θα σας έβρισκε αντίθετη μια τέτοια κίνηση του, του την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τα προϊόντα καπνού γίνεται λόγος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, για τα πουρα, για τις αρωματικές ε, ουσίες που έτσι κι αλλιώς τα πουρα δεν χρησιμοποιούνται, ε, και το γαπνό που χρησιμοποιείται σε ναργιλέδες και τέτοια προϊόντα. Έχετε να μας πείτε τίποτα σχετικά. Και επίσης, ε, μέχρι το 2025 ε, τι θα γίνεται με τα απορρίμματα, τα απόβλητα τροφίμων. Έχουμε μια νομοθεσία τώρα για την σήμανση των αυγών ε, και ο κόσμος αρχίζει και πετάει τα αυγά. Ε, εμείς έχουμε στη Σουηδία μια νομοθεσία που επιτρέπει να τα κρατάμε στο ψυγείο για τρεις εβδομάδες, ξέρω εγώ. Και μετά ξαφνικά αρχίζουν και τα πετάν. Τι θα κάνετε για να μειωθούν ε, τα απορρίμματα τροφίμων μέχρι το 2025. Θυμίζω ότι είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό μέσο. Αυτό θα έχει να κάνει με τη χρήση ε, φυτοφαρμάκων, τη χρήση γεών, ε, τα απόβλητα, τη διαχείριση των υδάτων, των λιμάτων. Ε, βοηθάει και για το περιβάλλον αλλά και για τις οικονομίες. Ανησυχώ και εγώ με τη Λίντα Μακάβεν εξίσου για τις κρεοσκοπήσεις και επιθεωρήσεις. Ότι θέλετε να δώσετε αυτές τις εξουσίες στις εταιρείες. Ανησυχώ. Και τελευταία ερώτηση για την πλήρη πληροφόρηση ε, για τη σήμανση προϊόντων υνοπνευματοδών. Ε, πώς θα το κάνετε, πώς θα προλάβετε, έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συνειδητοποιήσουν. Εντάξει, περισσότεροι ξέρουν ότι το ενόπνευμα μεθάει και να μην πίνει πολύ γιατί θα μεθύσεις. Αλλά πολύ λίγοι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά συμβάλλει το ενόπνευμα ε, στην παχυσαρκία, γιατί είναι βόμβα θερμίδων. Ευχαριστώ η κυρία Ρόσμπαχ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων είναι κάτι ε, που με ενδιαφέρει και θέλω να αναφέρω. Εδώ η νομοθεσία, ξέρετε, έχει έρθει πάρα πολύ αργά ε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ να νομοθετήσουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για ε, τις συσκευασίες ε, για τη χρήση φαρμάκων σε προϊόντα ζωικά ή μικροβιακά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να φέρει ένα κείμενο το συντομότερο. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Έχουμε πολλές εκθέσεις, ανακοινώσεις, συμπεράσματα που εκδόθηκαν και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και γιατί αναβάλλεται τώρα αυτό από προθεσμία σε προθεσμία, παρατείνεται συνεχώ. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, κύριε Επίτροπε, γιατί οι νομοθετικέ προτάσει δεν φτάνουν στο Κοινοβούλιο, τώρα που έχουμε ακόμα ευκαιρία να ε, περάσουν και με τρόπο σωστό. Και προλαβαίνουμε είναι ακόμα εφικτό αυτό στην παρούσα θητεία, αν έχουμε όμω την πολιτική βούληση. Θα πρέπει το συντομότερο να κατατεθούν αυτέ οι προτάσει. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για τη δημόσια υγεία γενικότερα. Ευχαριστώ. κυρία Λιωτάρ, τελευταία συντονίστρια. Ευχαριστώ κύριε Μπόρτ. Χαίρομαι που σα βλέπω εδώ και σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Είπατε ότι φαίνεται δύο προτάσει για την κλωνοποίηση και τα νέα τρόφιμα. Περιμένω να δω τι θα περιέχουν οι προτάσεις αυτές, πάντως χαίρομαι. Είπατε ότι θα μας μιλήσατε ε, για ε, τις ε, επιπτώσεις καθυστερημένες αυτές. Πότε όμως, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες, ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντική ε, αυτή η ρύθμιση και μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου. Θα πρέπει οι καταναλωτές να ξέρουν τι έχουν στο πιάτο τους, ε, είτε είναι ζήτημα ασφαλείας, είτε είναι ζήτημα ε, απάτης, αν τρώνε δηλαδή μοσχάρι, άλογο ή κλωνοποιημένο ζώο. Πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έχουν υπογράψει για ένα οχτάωρο ε, στη μέγιστη διάρκεια μεταφορά ζών των ζώων ε, που προορίζονται για σφαγή. Θα έρθει αυτή η πρόταση. Επιτέλους, γίνεται μεγάλη συζήτηση ε, για την μελέτη που έκανε η ΕΦΣΑ για τους κινδύνους από την Ασπαρτάμι. Και αυτό το θέμα είναι και πολιτικό και επιστημονικό. πρόσφατα έδειξαν στοιχεία ε, ε, οι ε, αρχές της Ιταλίας και της Γαλλίας, οι αρμόδιες, αντίστοιχο σε φέτα, πούμε, θέλουν να μειώσουν τα όρια προς τα κάτω πριν περιμένουν να έρθει η μελέτη της ΕΦΣΑ. τι λέτε γι' αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος για να απαντήσει σε ερωτήσεις των συντονιστών. Παρακαλώ. Για την πρώτη ερώτηση ο Λίζε για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εξοικονόμησης. Στις χώρες, από τις χώρες αυτές ορισμένες ε, προσήλθαν στα προγράμματα αυτά ε, ε θελουσίως, σε άλλες επευληθεί. Βέβαια είναι θέμα εμπειρίας. Αρχίζουμε τώρα και εμπλεκόμαστε ιδίως στις τελευταίες διασώσεις με συνοδευτικά προγράμματα, όχι βέβαια λιτότητα για τη λιτότητα, αλλά χρειάστηκε να λεφθούν μέτρα για να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα. Διότι αν δεν δώσουμε το φάρμακο, τότε η νόσος θα, ε, η ασθένεια δηλαδή θα επεκταθεί και θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη. Αλλά βέβαια η υγεία παραμένει ευθύνη δική τους. Η εισαγωγή μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη, δα, καλύτερη δαπάνηση των πόρων ε, με... και εγώ πήγα στην ε, Ελλάδα τον Φεβρουάριο που μας πέρασε όχι για να τους ελέγξω αλλά για να βοηθήσω ο ρόλος μου δεν είναι ο έλεγχος η Κομισιόν δεν μπορεί να παίξει το ρόλο των μη κρατικών οργανισμών. Εμείς έχουμε θεσμικό ρόλο, να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Εάν βέβαια δεν σέβονται το δίκαιο, τότε εμείς προσφεύγουμε εναντίον τους. Πάντως, καταρχήν, ο ρόλος της Κομισιόν να βοηθεί χώρες και κυρίως εκείνες που χρειάζονται το, τη βοήθεια. Παρά την κρίση και παρά τις δυσκολίες που υφίστανται και παρόλο που ακόμη δεν έχουν ξεφύγει από τα δύσκολα, έχουν ωστόσο ληφθεί ορισμένα μέτρα τα οποία περιόρισαν τα πάνε. Σας αναφέρω δύο. Η χρήση περισσότερων γενώσιμων φαρμάκων κατόρθωσε να μειώσει τις πραγματικά αστρονομικές στην Ελλάδα δαπάνες για φάρμακα. Και βεβαίως είδαμε τη Σουηδική κυβέρνηση να βοηθά την ελληνική κυβέρνηση για να εισαγάγει ένα σύστημα ηλεκτρονικών συνταγών που τώρα είναι από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη για τα φάρμακα κτλ. Βεβαίω υπάρχουν άλλα προβλήματα, δηλαδή της πρόσβασης του κοινού και των μη ασφαλισμένων εργατών που δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα. Και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά ας μην δίνουμε την εντύπωση ότι η Κομισιόν τα κάνει αυτά από ευχαρίστηση, δηλαδή παίρνει το πελέκι και κόβει το κόστος μόνο για χάρη της λιτότητας, όλα πρέπει να έχουν ένα σκόπο. Ε, σκοπός είναι δηλαδή η διάσωση του συστήματος. Βέβαια, εάν με ρωτήσετε αν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα σε κάποια επιδείνωση της υγείας και των δημοσιονομικών περικοπών, βεβαίως η απάντηση είναι ναι. Παρόλο που, εάν εξετάσει κανείς πάλι την Ελλάδα και δει την αύξηση του ρυθμού των αυτοκτονιών, αυτό δεν έχει σχέση βέβαια με την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας, αλλά περισσότερο με την δημοσιονομική κατάσταση, την οικονομική κατάσταση. Είδα στην Ελλάδα ότι υπάρχει και αύξηση του αριθμού των ε, προσώπων φορέων του ιού του AIDS. Η κυβέρνηση, η μου λέει ότι αυτό οφείλεται στην ε, μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ εξετάζω το πρακτικό, την πρακτική σκοπιά του θέματος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτό τον αυξανόμενο αριθμό των ε, φορέων HIV για τις επιθεωρήσεις και ιδίω όσον αφορά την υγιεινή. Θα υποβάλουμε πρόταση στο τρίτο τρίμηνο του έτους, όχι με το σκόπο να χαμηλώσουμε τις προδιαγραφές, αλλά να εντοπίσουμε σε ποιους τομείς είναι μεγαλύτερη κίνδυνη. Και βεβαίως το κρέας έχει μεγαλύτερους κινδύνους ρίσκο δηλαδή από ότι άλλα τρόφιμα και δεν θα αφήσουμε βέβαια το θέμα διότι θέλουμε να διατηρήσουμε την καλή μας φήμη και η καλή μας φήμη είναι ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει από τα καλύτερα συστήματα εξασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη συνέχιση των τεστ, είτε πρόκειται για αλόγου είτε πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων κλπ. Για το θέμα του κρέατος αλόγου, η αντίδραση των χωρών μελών ήταν πέραν πάσης προσδοκίας θετική. Για παράδειγμα του Ενωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα της Γερμανίας, αλλά και όλων των χωρών μελών. Αποφάσισαν δηλαδή να διεξαγάγουν τα τεστ αυτά, ακόμη και αν, παρόλο που, δεν ήταν παρά μόνο σύσταση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ πιστεύω ότι σε περιόδους προβλημάτων και κρίσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατάξει την εκτέλεση των τεστ αυτών, των ε, δοκιμασιών αυτών. Και αυτό θα μπει και στο νέο πακέτο το οποίο θα υποβάλουμε. Βέβαια, εφαρμόστηκαν πλήρως οι συστάσεις από τις χώρες μέλη και όσο γνωρίζετε εμείς δημοσιεύσαμε αμέσως και τα αποτελέσματα. Βέβαια, οι επιθεωρήσεις εξακολουθούν να είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όταν οι έλεγχοι έγιναν από, τα, από τις χώρες μέλη ήταν ακριβέστεροι από τους ελέγχους που, κάνουν οι, που κάνει ο ίδιος ο κλάδος. Προσοχή λοιπόν εδώ. Φαίνεται ότι οι έλεγχοι που διεξήγαγαν οι χώρες μέλη ήταν καλύτεροι από αυτούς που κάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που σας λέω τώρα δεν είναι δάπηχη προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι γεγονός. Για τις μέλισσες, κύριε Ντέιβις, εξεπλάγην από την αντίδραση των χωρών μελών. Πρώτη μου εμπειρία του είδους αυτού, διότι εγώ νόμιζα ότι επειδή η ΕΦΣΑ συνήθως επικρίνεται ότι δήθεν είναι πολύ χαλαρή και λέει ναι σε όλα, στην περίπτωση αυτή που είπε όχι, οι περισσότερες χώρες μέλη ανέμενα ότι θα δέχονταν την άποψη αυτή. Ωστόσο, διόλου ομαλό δεν ήταν το έδαφος, διότι παρόλο που υπήρχε επιστημονικά θεμελιωμένος αριθμός ενδείξεων, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έγιναν μελέτες επιτόπου, field studies, που να οδηγήσουν στην γνώμη της ΕΦΣΑ, που να λέει ότι όχι όλα τα νέα νοικοτινοειδή έχουν αυτές τις βλαβερές συνέπειες για τις μέλισσες, αλλά ορισμένα στοιχεία, ορισμένα, ιδίως τρία νέα νοικοτινοειδή, προκαλούν αυτό τον αποπροσανατολισμό των μέλισσων που οδηγεί στην εξάλληψη των αριθμών τους. Εγώ λοιπόν εξεπλάγιν διότι νόμιζα ότι οι περισσότερες χώρες μέλη θα δέχονταν την γνωμοδότηση αυτή. Άλλωστε δεν επρόκειτο παρά μόνο για αναστολή χρήσης για δύο χρόνια για να μπορέσει να μελετηθεί αν όντω έχουν αυτή την βλαβερή συνέπεια τα νοικοτινοειδή. Και ωστόσο υπήρξε ένας αριθμός ενστάσεων και ψήφων κατά. Τώρα πρέπει να πω βέβαια από την άλλη μεριά ότι ορισμένες χώρες μέλη ήδη είχαν εισαγάγει απαγορεύσεις χρήσης αυτών των ε, ε, φυτοφαρμάκων πριν από την σύσταση, τη γνωμοδέτηση και δεν αντιμετώπισαν τέτοιες αποκαλυπτικές εντό εισαγωγικών ε, καταστροφικές επιπτώσεις. Ορισμένες μάλιστα ήταν και κάποια αύξηση του αριθμού των πληθυσμών των μελισσών. Τώρα δεν είμαι δογματικός για να πω ότι δεν και καλά η μείωση του αριθμού των μελισσών οφείλεται μόνο χά στη χρήση αυτών των Ιζανιοκτώνων. Δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι ένας από τους παράγοντες, εκτός από την κλιματική αλλαγή, εκτός από τις ασθένειες, που οδηγούν στη μείωση του αριθμού των μελισσών, είναι και η χρήση ορισμένων ειδών νέων νικοτινοειδών Και επειδή είδαμε και στην Διαρκή Επιτροπή την θέση ότι, που τελικά οδήγησε στο να μην υπάρχει ειδική πλειοψηφία υπέρ της θέσης, παρόλο που υπήρχε πλειοψηφία των χωρών μελών και κατά τον αριθμό τους αλλά και κατά τη στάθμιση των ψήφων υπέρ της προτάσεως, εμείς μείναμε ακριβώς μέσα στα πλαίσια της νομοδότησης της ΕΦΣΑ με τις εξαιρέσεις για τα θερμοκήπια και για ορισμένες εσοδίες που δεν ορισμένες καλλιέργειες δηλαδή, που δεν ε, βλάπτουν τις μέλισσες, μπορεί να χρησιμοποιούνται μετά από την ανθοφορία και κάποιες χρήσεις που συζητούνται βέβαια στην ΕΦΣΑ ακόμα. Τώρα δύο χρόνια θα είναι αρκετά Αυτή ήταν και η απόφαση των χωρών μελών. Να αρχίσουμε δηλαδή με μια διετή περίοδο για να δούμε εάν όντως μπορούν να προκύψουν κάποια αποτελέσματα από τα τεστ αυτά και από την απαγόρευση. Λάβαμε τώρα και ειδήσει ότι υπάρχουν και άλλα ζυζανιοκτώνα τα οποία των οποίων επιτρέπεται η χρήση, αλλά έχουν και αυτά τις ίδιες βλαβερές συνέπειες για τις μέλισσες. Εφόσον αποδειχθεί αυτό, θα επανέλθω για το θέμα αυτό, γιατί είναι βέβαια σημαντικό να προστατευτούν οι αριθμοί των μέλισσών και βεβαίως να ενημερωθεί και το κοινό για την σημασία των μελισσών. Σε ορισμένες χώρες μαθαίνω ότι πηγαίνουν οι άνθρωποι τώρα και γονιμοποιούν τα ε, φυτά με το χέρι, διότι δεν υπάρχουν πια οι μέλησες. Σε αυτό το βαθμό έχει φτάσει η κατάσταση. Και μάλιστα τώρα προσφεύγουν και ορισμένες εταιρείες κατά των αρχών που έχουν επιτρέψει τη χρήση των, των ε, αυτών. Ναι, θα παρακολουθούμε λοιπόν την δράση των χωρών μελών για την εφαρμογή της απαγόρευσης καλλιντικών που έχουν παραχθεί με χρήση πειραματοζών και βέβαια να βάλουμε κάποια τάξη ε, ε, από την άποψη αυτή. για τα πουρα, τα τσιγαράκια, τα πουράκια, τις αρωματικές ουσίες. Υπάρχει μια πρόνοια στην οδηγία για τον καπνό που λέγει ότι δεν θα τα ρυθμίσουμε αυτά, τις αρωματικές ουσίες και τις γεύσεις και τα λοιπά, εκτός αν δείξουν οι στατιστικές ότι αυξάνεται η κατανάλωση των προϊόντων αυτών. Δηλαδή, εάν αργότερα φανεί ότι τα προϊόντα αυτά που είναι πολύ περιορισμένα στην κατανάλωσή τους ε, δείξουν αυξημένη κατανάλωση ακριβώς γιατί εξαιρούνται από κάποιες διατάξεις και πρόνοιες της οδηγίας, τότε μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες ρυθμίσεις για τα προϊόντα αυτά και για τα προϊόντα. Δηλαδή δεν έχουν εξαιρεθεί απολύτως ε, από το πεδίο εφαρμογής ε, του κανονισμού αυτού. Αναφέρονται στη ρύθμιση. Λοιπόν, για την κλωνοποίηση, μάλιστα, περιμένουμε τη μελέτη αντικτύπου και την αντίστοιχη έκθεση που θα κατατεθεί. Ελπίζω να νομοθετήσουμε, γιατί βρισκόμαστε τώρα στην εξή περίεργη κατάσταση. παραμένει ακόμα δυνατή ε, η κλωνοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνικά, έτσι, νομικά. Ξέρω ότι γίνεται γενικά συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και εκτός του Κοινοβουλίου ε, ε για την επισήμανση. Αλλά πώς θα γίνει αυτό σε περίπτωση ε, που υπάρχουν κλωνοποιημένα ζώα. Ξέρουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και θα πρέπει να προτείνουμε μία λύση για να έχουμε κάποιο είδου νομοθεσία και από αυτού του θέματος. Πιστέψτε με ότι είναι δύσκολο καμιά φορά να δρομολογήσει κανείς ε, κάποιες ε, νομοθετικές προτάσεις. Να ξεκινήσει δηλαδή η προσπάθεια. Ποια θα ήταν η τραγωδία να προχωρήσουμε σε εκτενή νομοθεσία χωρίς να έχουμε τα στοιχειώδη. Δηλαδή, όταν φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της, θα πρέπει να ξέρει ποιε είναι οι πιθανότητες να εγκριθούν από τους συνομιθέτες οι προτάσεις. Αν είναι προφανέστατο ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί η νομοθεσία, τότε καλύτερα να αφαιρώσουμε το χρόνο μας σε άλλα θέματα ε, που ε, έχουν πιθανότητες να περάσουν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ή σε ένα εύλογο χρόνο για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει έρθει μια πρόταση. Ε, ολοκληρώνεται αυτό το καιρό ε, στο Συμβούλιο για τη μελέτη αντικτύπου για να βρούμε τη σωστή ε, πρόταση και ισορροπία για τα ε, αντιβιωτικά που αντέχουν τα μικρόβια σε αυτά θα πρέπει να ε, διατηρούνται για ανθρώπινη χρήση και ποτέ για ακτινιατρική χρήση. Σε ό,τι αφορά τη σήμανση των ινοπνευματοδών, μάλιστα περιμένουμε ε, αξιολόγηση της στρατηγικής για το ινόπνευμα και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα μέχρι τα τέλη του έτους. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, ακολουθεί ο επόμενος γύρος τώρα συναδέλφων, ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Χάρηκα πάρα πολύ ως συμβατικός αγρότης που ήσασταν σκληροί στην αντιμετώπιση αυτών των φυτοφαρμάκων. Το θέμα δεν είναι ότι έχουν οι μέλισσες τόσο καλό λόμπι. Αλλά το θέμα πάει πολύ πιο βαθιά από τις μέλισσες και τα λόμπι. Πρέπει να σας πω ότι στη δική μου περιφέρεια τα έντομα ε, και οι πολύ μικροί οργανισμοί κινδυνεύουν πηγαίνετε στον κάτω ρήνο χωρίς να καθαρίσετε δύο εβδομάδες το αυτοκίνητό σας να το πλύνετε, δεν θα υπάρχει ούτε μιγάκι στο παρμπρίζ. Ε, μια φορά το χρόνο ψεκάζαμε, ραντίζαμε, ε, φεύγαν τα έντομα και μετά ξαναρχόντουσαν. Τώρα έχουμε συνεχείς ψεκασμούς και ραντίζουμε πραγματικά έστω και συμβατικός αγρότης ε, που μπορεί να είμαι, δεν το καταλαβαίνουν οι συμβατικοί αγρότες, αλλά θα το μετανιώσουν πικρά. Διετία δεν είναι τίποτα. Παρακαλώ να το διπλασιάσετε και πολύ εντατικά, επιστημονικά και τελείω νυφάλαια και ψυχρά να τα ελέγξετε όλα αυτά. Έρχομαι τώρα στα προϊόντα καπνού. Δεν θα μιλήσω ούτε για πακέτα τσιγάρων, ούτε για πουρα, ούτε για τίποτα τέτοιο. Θέλω να πω το εξή. Έγινε μεγάλη μάχη, καυγάς ομυρικός και αποφασίσαμε ε, ότι θα πρέπει στο REACH να ελέγχονται και τα προϊόντα καπνού από τη βιομηχανία. Το είχαν σημειώσει πάρα πολύ και είπαν όχι είναι φυσικό προϊόν ο καπνός, άρα εξαιρείται από το REACH. Ναι, αλλά ε, δεν είναι ο καπνός ε, φυσικό προϊόν όταν αναμειγνύεται με 50-60 χημικές ουσίες που το γνωρίζουμε. Ξέρω ότι εσείς δεν είστε αρμόδιο για το ΡΙΤΣ, αλλά σας λέγω ότι πραγματικά η καπνοβιομηχανία εκφεύγει των ευθυνών τη. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Ε, ε, ε υπάρχει... Ε, όχι τρύπα στο φράχτη, φράχτη στην τρύπα. Είναι τεράστια η τρύπα και φεύγει η μηχανή. Λοιπόν, είπαμε 1,5 λεπτό, δεν είναι ε, Η κυρία Ροτμπέρεν, συμφωνώ απολύτω με τον ε, κύριο Φλόρενς. Ευχαριστώ που ήρθατε, Επίτροπε. Μερικές ερωτήσεις. Πέντε προτάσεις ε, καταθέσατε χτες για να αντικαταστήσουν 70 νομοθετικές προηγούμενες. Μήπως χάσατε την ευκαιρία να επαναφέρετε την ιδέα σήμαση για τη χώρα προέλευσης για όλα τα προϊόντα κρέατος δεν είναι απαραίτητο ε, ένα θέμα ε, ασφάλειας ανθρώπινας υγείας ή δημόσιας υγείας. Είναι θέμα όμως προστασίας του καταναλωτή, ενημέρωσης του καταναλωτή, καταπολέμηση της απάτης και εμπορίου. Θα πρέπει να δράξετε αυτή την ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές συσκευές και ε, μηχανήματα γενικότερα. Ε, δεν ξέρω εάν είναι ευφυής η ιδέα να αφαιθεί στα χέρια κάποιου που θα αναλάβει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω, δεν το κρίνω. Ε, λέτε ότι αυτή η πρόταση θα ε, εμποδίσει την καινοτομία. Ναι, δεν, το ξέρω, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε την καινοτομία γιατί χρειαζόμαστε απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να προστατεύουμε και τους ασθενείς. Ε, ξέρετε τι έγινε με τα εμφυτεύματα ε, κεφαλής ή υγοφού χωρίς ελέγχους, χωρίς ε, σωστή αντιμετώπιση. Ε, πιστεύετε πραγματικά ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός ελέγχου πριν κυκλοφορήσει ένα προϊόν στην αγορά, μετά που θα κυκλοφορήσει, μήπως χρειάζεται κάποια διαφορετική μορφή αδειοδότησης γενικότερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεπάζ για μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Πρώτον, συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ για την προέλευση, τη γεωγραφική προέλευση του κρέατος. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ έχουν μια τέτοια απέτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμεί δεν το κάνουμε όμω. Δεύτερον, κύριε Επίτροπε, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η απάντηση η οποία δώσατε στην κυρία Διωτάρ όσον αφορά το ζήτημα τη κλωνοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με ξεκάθαρο τρόπο 2008 και απέρριψε τη χρησιμοποίηση της κλωνοποίησης. Και αυτό το που μας είπατε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την κλωνοποίηση αρκεί να υπάρχει μια επισήμανση. Και μας λέτε ότι η κλωνοποίηση αδειοδοτείται, δεν υπάρχουν κανόνες βέβαια και έχετε δίκιο προς αυτό, και ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές, το γνωρίζετε όμως αυτό, δεν θέλουν να τρώνε κλωνοποιημένο κρέας και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή είναι πραγματικά απαράδεκτη. Επομένως, κύριε Επίτροπε, τι μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον προσωρινά, τουλάχιστον για να πούμε προς τον Ευρωπαίο καταναλωτή ότι μπορεί να επιλέγει σωστά το κρέας και ότι μπορεί να αποφύγει το κλωνοποιημένο κρέας. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού πρέπει να λάβει πολύ γρήγορα δράση. Ως προς την Ασπαρτάμι τώρα. Έγινε μία συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχε εκπρόσωπος της ΕΦΣΑ και της DG Sanko, όπου η έκθεση της ΕΦΣΑ για την Ασπαρτάμι επικρίθηκε πάρα πολύ και τέθη αμφιβόλο αμφιβόλω μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σας η στάση και τι πρόκειται να κάνετε για τη σχετική ρύθμιση όσον αφορά την Ασπαρτάμι δηλαδή. Ευχαριστώ κυρία Ριβαζή για μισό λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε επίτροπε που ήρθατε στην συνεδρίασή μας, μας δίνετε πάρα πολλές πληροφορίες και απαντάτε και σε κάποιες από τις ανησυχίες μας. Τώρα, όσον αφορά τα ενδοκρινικά, ε, τις ενδοκρινικές δοκιμές οι οποίες γίνονται, πληροφορίες που μας είχαν δοθεί αρχικά από την ΕΦΣΑ και από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όσον αφορά στοιχεία όπως τα παραμπέν για παράδειγμα. Στις δοκιμές λοιπόν αυτές που έχουν γίνει, γιατί ξέρετε κάθε φορά που θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι ενδοκρονικές παθήσεις που μπορούν να προκύψουν από τα καλλιντικά, ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε κάποιες ε, χημικές ουσίες οι οποίες επηρεάζουν τον καταναλωτή, αναφέρουμε στους ενδοκρινικούς διαταρακτές, όχι τόσο ως προς την ποσότητα, αλλά ως προς την έκθεση, την ίδια την έκθεση των καταναλωτών στους ουσίες αυτές. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταρακτές. Τώρα, όσον αφορά τις ιατρικές συσκευές, ξέρουμε ότι έγινε μια συνεδρίαση για το ζήτημα αυτό και ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο στη Μασαλία με εμφυτεύματα καθώς επίσης και ένα σκάνδαλο με τα εμφυτεύματα κεφαλής μυριαίου. Θεωρώ ότι αν είχαμε μια πιο αυστηρή νομοθεσία για τα εμφυτεύματα δεν θα είχαμε τα σκάνδαλα αυτά με τα εμφυτεύματα τα οποία είχαν δώσει κάποιες, κάποια νοσοκομεία σε ασθενείς. Επίσης, ξέρετε ότι η ΑΠΒΗ, μία φαρμακοβιομηχανία, είχε ταχθεί κατά τις αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φάρμακα όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές που είχαν γίνει. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να υπάρχει πρόσβαση στις κλινικές δοκιμές. Αν όμως επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, τότε οι φαρμακοβιομηχανίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα κάθε φορά να επισύρουν στο δικαστήριο την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Ρεμπέκα Τέιλορ. Ε, μια σύντομη ερώτηση. Σίγουρα θα γνωρίζει ο Επίτροπος ε, ε, ότι ε, έγινε μια προσφυγή κατά της απόφασης της σκοτικής κυβέρνησης για την ελάχιστη τιμή στα πνευματο δι, ποτά. Ξέρετε ότι αυτή η προσφυγή να βάγισε. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. ο Ζιλ Παρνιό, παρακαλώ. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να σας πω ότι χτες το βράδυ, όπως θύμισε ο πρόεδρος, συμφωνήσαμε στον τριμερή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλανδική Προεδρία σε ό,τι αφορά τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Ε, θέλουμε να συζητηθεί και να ψηφιστεί αυτή η πρόταση κατά την Ολομέλεια του Ιουνίου φέτος, διότι θεωρώ ότι το θέμα είναι πήγον. Αν δούμε τι γίνεται στην Κίνα με ε, το στέλεχος του ιού ή τα 7 νη 9 που σήμερα ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες θα ήθελα να χαιρετήσω γιατί κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου πρωτοστάτησαν και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ πραγματικά ε, υπήρξε ε, διαμεσολαβητής. Λοιπόν, αυτός ο ιός είναι κάτι που μας ανησυχεί και θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη και πού βρισκόμαστε ως προς την εξέλιξή του. Γνωρίζουμε ότι τελικά μπορεί να υπάρξει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. 25% ήδη των περιστατικών που δυστυχώς, δυστυχώς κατέληξαν 11 ημέρες μετά τη δήλωση, την εκδήλωση μάλλον της ασθένειας. Και βλέπουμε και μετάλλαξη του στελέχους του ιού. Ένα δεύτερο η βυσφενόλη α. Ε, ε, ζητήσαμε, αποτινεύσα μια μελέτη και η οποία ανέβαλε ε, το πόρισμα. Ενώ στη Γαλλία ασχολούνται 200 ερευνητέ με αυτό, έχουν μελετήσει την ουσία τη φαινόλη α και έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνα. Εσείς τι λέτε για όλο αυτό. Ευχαριστώ Κύριε Ακονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα ενώπιον μας για άλλη μια φορά για να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχω δύο ερωτήσεις εγώ. Σύντομα. Η μία ιδιαιτέθη είναι για το κλωνοποιημένο κρέας. Αυτό τον καιρό εξετάζουμε μια έκθεση που αφορά ένα κανονισμό για την ηλεκτρονική σήμανση των βοηδών ε, και του, συνέχεια την επισήμανση, την ετικέτα στο κρέας τους. Υπάρχει αυτό το θέμα του κλωνοποιημένου κρέατος, μάλλον κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα. Μας είπατε ότι τον Ιούνιο του 2013 θα φέρνατε πρόταση. Σας είχα ρωτήσει και μάλιστα αυτά τα δηλώσατε στις 13 Νοεμβρίου του 2012. Ξέρω ότι απαντήσατε αλλά ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Δεύτερον, κατά την πρόταση του νομοθετικού πακέτου μας είπατε ότι περιμένετε ε, μια μελέτη αντικτύπου ως προς το βόλιο κρέας, ε, το ε, κρέας αλόγου και τις σχέσεις τους με τα προϊόντα κρέατος μετά την επεξεργασία. Τι θα γίνει με αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θα έρθει πριν τα τέλη του έτους. Τώρα που βρισκόμαστε, θα την έχουμε στη διάθεσή μας εγκαίρως. Εγώ παρακολουθώ τον κανονισμό της επισήμανσης του βοήου κρέατος και θα ήθελα κύριε Επίτροπε να μας πείτε εάν μπορούμε να επωφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας για να εντάξουμε στον παρόντο κανονισμό μια αντίστοιχη τροπολογία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Όσον αφορά τους πόρους, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, αφού βέβαια μελετήσουμε πρώτα την πρότασή σας κύριε Επίτροπε, σε κάθε λεπτομέρεια. Σήμερα θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω εσάς κύριε Επίτροπε, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες της DG Sanko για την εργασία που έχετε καταβάλει όσον αφορά την ε, αναστολή της χρησιμοποίησης των ε, νεονικοτινοειδών αυτών Ξέρω ότι δεν ήταν ε, εύκολο, δεν ήταν εύκολο το έργο σας, ούτε ήταν εύκολο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα πάντως να σας θέσω δύο επιμέρους ε, ερωτήσεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις μέλησες και τα ζενεοκτώνα. Πρώτον, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ανέστηται τη χρήση τριών νέων νοικοτινοειδών, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο νέο νοικοτινοειδές το οποίο αδειοδοτήθηκε, το φλόρ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια προθεσμία προβλέπετε προκειμένου να γίνει μια αξιολόγηση της ΕΦΣΑ για τα νέα αυτά νεονικοτινοειδή προϊόντα και για τα νευροτοξικά αυτά νευροτοξίες ουσίες προβλέπονται και έπειτα όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι. Για ποιο λόγο σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει ακόμα αξιολόγηση αντικτύπου, προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο και πότε. Ευχαριστώ. Κούκοβιτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία και η υγεία των τροφίμων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, άλλο συμπληρώνονται. Επομένως, το Ινστιτούτο της Σλοβενίας ξεκίνησε ένα, μια έρευνα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος της μελέτης αυτής είναι να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση τοπικών και υγιεινών τροφίμων και να ενθαρρύνει ουσιαστικά τη χρησιμοποίηση λαχανικών και άλλων ε, τροφίμων στα πλαίσια μιας υγιεινούς διατροφής, στοιχεία της διατροφής μας τα οποία έχουμε ξεχάσει και τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε. Δύο ερωτήσει λοιπόν θα ήθελα να θέσω. Η υγεία προφανώ εξαρτάται πάρα πολύ από τα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει συγκεκριμένε μελέτε στον τομέα αυτό. Και ποια είναι, η σημα... ποια είναι τα πορίσματα των μελετών αυτών. Δεύτερον, έχουμε εξετάσει τον αντίκτυπο στην υγεία και για αυτέ τι τέσσερι μορφέ ε, τροφό όσον αφορά για παράδειγμα τα λαχανικά, όσον αφορά το σκόρδο ή και άλλε τροφές που δεν χρησιμοποιούμε τόσο συχνά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι απαντήσει που ήδη δώσατε όσον αφορά του σπόρου. Εντίτε Στρέλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μία ερώτηση έχω να κάνω όσον αφορά την αύξηση ανισότητας για την υγειονομική περίθαλψη στα κράτη-μέλη. Το 2009 Ευρωπαϊκή Επίτροπη σε μία ανακοίνωσή της όσον αφορά την ισότητα στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση των υγειονομικών τη υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για την οποία εγώ ήμουν εισηγήτρια, μας είχε πει ότι θα παρουσίαζε μια ενδιάμεση έκθεση όσον αφορά την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον τομέα αυτό ήδη από το 2012. Δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα την ανακοίνωση αυτή, μόλον ότι είμαστε πια στο 2013. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί έκτοτε σε πάρα πολλά κράτη-μέλη, ιδίως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Κύπρο και στην Ισπανία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Γνωρίζετε ότι έχει επέλθει μια επιδείνωση όσον αφορά την ισότητα πρόσβασης στις ε, στην υγειονομική περίθαλψη στις χώρες της λεγόμενης διάσωσης και αν ναι, ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει προκειμένου να μειωθεί αυτή η ανισότητα στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάνει επίση μια γενικότερη εξολόγηση του αντικτύπου των μέτρων λιτότητα στι χώρε αυτέ στον τομέα τη υγεία. Ευχαριστώ, κυρία Κάντεμπαχ. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο ε, για τη συνέπειά του, για την επιμονή του, για τα νεονικοτινοειδή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορώ να συμφωνήσω παρά να συμφωνήσω με τον Χάιντς Φλόρεντς είναι ένα από τα θέματα, απομένουν πολλά ακόμα ανοιχτά και θέλω να αναφερθώ και σε αυτά. Είπατε κι εσείς ότι δεν είναι μόνο τα φυτοφάρμακα, είναι θέμα και της βιοπικιλότητας. Θα πρέπει να ε, παραμείνουν ε, στη φύση τα έντομα που συμβάλλουν ε, στην επικονίαση. Σε αυτή την ιστορία με το πολλαπλασιαστικό υλικό του σπόρους δεν συμμεριζόμαστε το δικό σας ενθουσιασμό. Πραγματικά Περιορίζεται η ελεύθερη ανταλλαγή και κυκλοφορία εμπορευμάτων με το παλιό πολλαπλασιαστικό υλικό, το παραδοσιακό. Ε, ε, σας παρακαλώ να δείξετε συνέπεια όμως και στη βιοπικιλότητα και ε, στα έντομα της επικονίασης και για τους σπόρους, γιατί στο μεταξύ έχουμε αρκετές επιστημονικές αποδείξεις ότι γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό μειώνει την ποικιλότητα των ειδών και επηρεάζει αρνητικά και τα έντομα που συμμετέχουν στην επικονίαση και όταν πρόκειται για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τα θέματα υγείας αλλά και τα θέματα διατήρησης της ποικιλότητα των ειδών. Ευχαριστώ. Για αυτό που είπατε και που ζήτησε η Ντάκμα για την ε, ε, προέλευση, χτες ξεχάσαμε να το ζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ε, σας ε, ενθαρρύνω να ε, δείξετε την ίδια επιμονή και συνέπεια και στην διατήρηση των ειδών. Ωραία. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Θα θέλω να δώσω την ευκαιρία στον Επίτροπο να απαντήσει σε ερωτήσεις που έγιναν ή δυνατόν στο σύντομο χρόνο που μας απομένει. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ε, ερωτήσεις για την επισήμανση για το θέμα της χώρας προέλευσης. Όταν συζητήσαμε για το κρέας αλόγου, σας είπα ότι είμαι ανοιχτός να συζητήσω ό,τι θέλετε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Περιμένουμε ακόμα τη μελέτη αντικτύπου. Κανονικά επρόκειτο να κατατεθεί στα τέλη του έτους. Ε, προσπαθούμε να έρθει στα τέλη του θέρους αρχές φθινοπόρου και πιέζουμε και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα κάνουμε και τις προτάσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα και εσωτερικά και εσωτερικά πάντως υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες αλλά και βουλευτές όλο και περισσότεροι που πιέζουν υπέρ της πρότασης αυτής και στο Συμβούλιο αυξάνεται ο αριθμό των κρατών που θέλουν τη σήμανση αυτή την ετικέτα ε, για τη χώρα προέλευση. Βέβαια, τι εστί ε, χώρα προέλευση, που γεννήθηκε το ζώο, που εσφάγει το ζώο, ε, που έγινε επεξεργασία. Και υπάρχει ένα κόστο για όλη αυτή την ιστορία τη σήμανση. Και εγώ χαίρομαι για αυτό που είπατε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι τεχνικά αυτό δεν συνδέεται με το σκάνδαλο για το κρέας αλόγου, αλλά αυτή η ιστορία και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου έτσι πυροδότησε ακόμα περισσότερο ε, αυτή την πίεση. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε όμως και τι είδου σήμανση θα είναι αυτή η ετικέτα για τη χώρα προέλευσης. Αυτό αφορά για μη επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος. Ε, ε, το συζητάει το θέμα αυτό ο Επίτροπος Γεωργίας. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η σήμαση και θα πρέπει ε, το ε, προϊόντα κρέατος να έχουν ε, εναρμονισμένη ετικέτα με τα προϊόντα κρέατος που δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. Αλλιώς θα υπάρξει σύγχυση από νομικής πλευράς. Ε, εγώ είμαι πρόθυμος να συζητήσω ό,τι θέλετε για αυτό το θέμα. Και όσο περισσότερα είναι εκείνα τα κράτη που θέλουν να επιβληθεί αυτή η επισήμανση, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει η πρόταση. Γι' αυτό επιμένουμε εμείς στο χρονικό πλαίσιο, θέλουμε μάλιστα να ε, γίνουν οι προτάσεις λιγότερο ε, νωρίτερα, συγγνώμη. Ε, δεν θα έπρεπε να βγει όμως στη δέσμη μέτρων για την υγεία των ζώων είπαμε αρχές φθινοπόρου αντί τέλη του έτους να έρθει η έκθεση, η μελέτη αντικτύπου και μέχρι το 2014, τα τέλη του 2014 θα έχουμε. και την αντίστοιχη μελέτη αντικτύπου για άλλα προϊόντα ε, άλλων ζωικών ειδών, εγωπροβάτων, πουλερικών κτλ. Ε, μπορώ να δεσμευτώ προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά πάντα θα εξαρτηθεί από ε, κάποιες δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν. Πάντα υπάρχει ένα γραφειοκρατικό κόστος, ε, μια επιβάρυνση, ε, λογική όμως που θα πρέπει κανένας να αναβάνει αν θέλει μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ευχαριστώ για τα όσα είπε ο κύριος ε, Φλόρενς για τις μέλισσες. Η προστασία των αρουραίων ε, ίσως είναι πιο δύσκολη από την προστασία των μελισσών. Ε, γιατί οι μέλισσε είναι πιο δημοφιλείς από ότι τα ποντίκια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν ρόλο να παίξουν στη γεωργία και τα τροκτικά. Αναφερθήκατε στην ε, οδηγία ε, για τα προϊόντα καπνού, το λόμπι, την καπνοβιομηχανία. Κάτι που είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου θα ήθελα παρακαλώ να επαναλάβω. Όσοι είναι κατά των προτάσεών μας στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού, και αντίθετη στις δικές τροπολογίες, γιατί εσείς προσπαθείτε να είστε ακόμα πιο αυστηροί, όσοι λοιπόν διαφωνούν, δεν θα πούνε όχι ευθέως. Θα προσπαθήσουν να κολλησιεργήσουν, να επιβραδύνουν τη διαδικασία. Υπάρχουν τέτοιες απόπειρε. Ακόμα και για το ποιο σχηματισμό του Συμβουλίου θα πρέπει να το συζητήσει αυτό. Οι Υπουργοί Υγείας ή μήπως και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη γενική συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, όπου οι Υπουργοί Ανταγωνιστικότητας έχουν βέβαια διαφορετική στάση από τους Υπουργούς Υγείας. Μα αυτό είναι εξόχως ζήτημα δημόσιας υγείας. Αν καταφέρουμε να μειώσουμε έστω και κατά 2% τον αριθμό των καπνιστών, που σημαίνει 2,4 εκατομμύρια καπνιστές λιγότεροι, αυτό θα έχει και οικονομικές συνέπειες. Άλλες θα είναι ε, θετικές, άλλες αρνητικές. Τι πρέπει να κάνει ο Επίτροπος ε, της Υγείας στην Ένωση, να προωθεί το κάπνισμα για να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας ή να προστατεύει την υγεία του πληθυσμού. Και είναι και ρητορικό πολύ στο ερώτημα, διότι περιέχει την απάντηση. To ε, ε, για να είμαστε λοιπόν έτσι σόφρονες και προσεκτικοί, να μην αφήνουμε έδαφος εκείνους που δεν λένε ευθέω όχι, αλλά προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Ε, θα έρθει νέο κοινοβούλιο, θα οριστούν νέοι ε, εισηγητές, θα χάσουμε άλλη μια τριετία, ακόμα και όταν όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά και δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Αν χάσουμε τώρα την ευκαιρία να περάσει κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας, τα πάντα θα αναβληθούν κατά τρία ή τέσσερα χρόνια που είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Για το πολλαπλασιαστικό υλικό, του σπόρους, κυρία Κάντεμπαχ. Εγώ προσπάθησα να περιγράψω τα πραγματικά γεγονότα. Έχω μια φιλολογία και διαδίδεται αυτό και ε, στους βουλευτές και στους επιτρόπους. Αυτά δεν ευσταθούν. Πάντα μπορούμε να κάνουμε νομοθεσία για να διασκεδάσουμε τις φόβους και τις ανησυχίες ορισμένων που ανησυχούν για το τι κάνουμε. Μα το αντίθετο. Τα μέτρα ε, που προτείνουμε απελευθερώνουν ε, μια αγορά που είναι πάρα πολύ κλειστή και ελεγχόμενη σήμερα και για τους παραδοσιακούς πόρους. Εγώ με χαρά να δω όλες τις τροπολογίες σας για αυτό το θέμα και των συνομοθετών. Δεν ήταν καθόλου πρόθεσή μας Νομίζω ότι σας εξήγησα, εάν κάτι ξέχασα παρακαλώ να μου το πείτε. Δεν είναι καθόλου πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κανένα τρόπο να εμποδίσει το παραδοσιακό πολλαπλασιαστικό υλικό. Και τώρα κάποιοι πολιτικοί βγαίνουν και λένε ωραία πιέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλαξε θέση. Δεν ισχύει αυτό. Η θέση μας στην νομοθετική πρόταση ήταν πάντα ίδια. τροφή και σχέση της με την υγεία. Βεβαίως, τα χρόνια νοσήματα συνδέονται με την ε, έλλειψη σημαντικής άσκησης, ε, δεύτερο είναι η διατροφή, ε, κάπνισμα και ενόπνευμα. Αυτά τα τέσσερα. Και το συνδέω με το ενόπνευμα που με ρωτήσατε για το θέμα της σκοτίας και στην ελάχιστη τιμή των ενόπνευματοδών. Όλες οι μελέτες, τις οποίες γνωρίζω, και αφορούν μέτρα ελέγχου είτε του καπνίσματος είτε των υλοπνευματοδών έχουν αποδείξει ότι αντίθετα με τη λαϊκή πεποίθηση τα πιο αποτελεσματικά μέτρα είναι τα φορολογικά. Μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι εκστρατεία συνειδητοποίησης κατά του καπνίσματος ή κατά του υνοπνεύματος. Όχι. Εξεπλάγεν και ο ίδιος όταν έμαθα ότι τα φορολογικά μέτρα είναι εκείνα που πιάνουν τόπο. Άρα δεν είναι σωστό να λέμε ότι όταν αυξάνεται η τιμή του ινοπνεύματος ή των προϊόντων καπνού, τότε οι καπνιστές θα συνεχίσουν να καπνίζουν. Ή με τον ίδιο τρόπο όπως κάπνιζαν. Έχει αντίκτυπο. Μπορείτε να το θεωρήσετε ανάλγητο αυτό το μέτρο ή ομό ή οτιδήποτε, αλλά ε, πιάνει τόπο. Όσο αυξάνονται οι τιμές, το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα. Ε, όσο αυξάνονται οι τιμές των ε, ανθιγεινών τροφίμων, τόσο θα μειωθεί η κατανάλωσή τους. Χαίρομαι λοιπόν που οι σκοτικές αρχές εκέρδισαν αυτή την προσφυγή στα δικαστήρια εναντίον τους, δηλαδή απερίφθη. δεν θέλουμε να μην ευδοκιμούν τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τη συνθήκη και που βοηθούν στη μείωση κατανάλωση υνοπνευματοδών. Ε, Αν κοιτάξετε το προσδόκιμο ζωής ε, στην Ευρώπη, διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις συνήθειες και την κατανάλωση. Και είπα στους Υπουργούς Υγείας ότι Δεν έχει νόημα να διαμαρτυρόμαστε ε, για ε, τις δημοσιονομικές περικοπές. Ήδη έχουν επέλθει και έχουν πλήξει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχει δεχτεί περικοπή στον προπολογισμό της. Αντί λοιπόν να ε, διαμαρτυρόμεθα και να προσπαθούμε να αντιταχθούμε σε δημοσιονομικές περικοπές που έτσι καλλιώς θα επέλθουν, πιο εύκολο είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε. και να σχεδιάσουμε ε, με τέτοιο τρόπο τις περικοπές μας, ώστε να δαπανούμε λιγότερα χρήματα, αλλά παρόλα αυτά να διατηρούμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ε, φροντίδας υγείας και περίθαλψης. Τώρα, οι περικοπές στον προπολογισμό έχουν αντίκτυπο στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς. Η ψυχική υγεία, ας πούμε, σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχει επιπτώσεις λόγω της κρίσης της ίδιας, όχι λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε χάσει την κοινωνική μας πηξίδα πάντως, τουλάχιστον στην Επιτροπή και στην ε, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών, σε καμία περίπτωση και θα παρακολουθούμε την κατάσταση και σε αυτό. Όπως, σας είπα, όπως είπα και στην επίσκεψή μου στην Ελλάδα, ότι εμείς ήρθαμε να βοηθήσουμε, όχι να επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας, αλλά για να μπορούν βιώσιμα τα συστήματα υγείας, όλες οι χώρες, είτε είναι σε μνημόνιο είτε όχι, θα πρέπει να εισαγάγουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Το θετικό ποιο είναι. Υπάρχουν μέσα σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ε, δαπανούμε λιγότερα, αλλά να έχουμε κάποιες ε, στοιχειώδεις προδιαγραφές. Την άλλη εβδομάδα θα πάω στη Βόρεια Ιρλανδία για να κοιτάξω το σύστημα ηλεκτρονικής υγείας πώς εφαρμόζεται εκεί. Ε, έχουν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο σύστημα με 20.000 ασθενείς που συμμετέχουν και δεν είναι καν χώρα η Βόρεια Ιρλανδία, είναι περιφέρεια. Κοιτάξτε τι έκανε μία περιφέρεια. Θαύματα στα συστήματα αυτά. Ο κύριος Πεμιό ε, μίλησε για τους διασυνορικούς κινδύνους και απειλές για τη δημόσια υγεία. Χαίρομαι που τα αναφέρετε αυτά και ξέρετε και πολύ καλά το θέμα, ανησυχούσα εγώ πριν την έγκριση της οδηγίας αυτής από τον τριμερή διάλογο, διότι η αρχή της επικουρικότητας είναι ένα βολικό επιχείρημα και χρησιμοποιείται συνήθως για να αποτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχουν σε κάποια δράση. Σου λένε κάτω τα χέρια, αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Και για θέματα υγείας, η αρχή της επικουρικότητας είναι ακόμα πιο ισχυρό από ό,τι για άλλα θέματα. Και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω. Δύο φορές το χρόνο συναντιούνται μόνο οι Υπουργοί Υγεία, σε αντίθεση με άλλους σχηματισμού, όπως είναι η Γεωργίας κτλ. Εγώ θα προτιμούσα ένα τετράμινο, όχι ένα εξάμινο. Έχουμε τόσα θέματα ε, κλινικές δοκιμές, ε, οδηγία για τα προϊόντα καπνού, ιατρικές συσκευές. Πώς περιμένετε να αποφασίσουν για όλα αυτά τα θέματα οι ε, Υπουργοί Υγείας σε δύο ετησίως συνεδριάσεις, ένα εξάμεινο. Και είναι και τα άλλα θέματα, τα μη νομοθετικά που πρέπει να αποφασίσουν. Λέγω λοιπόν στους Υπουργούς Υγείας, η αρχή της επικουρικότητας έχει και άλλη όψη. Όχι μόνο τη μία, εμείς μόνο τη μία όψη αναφέρουμε, ότι δεν ανακατευόμαστε στα κράτη-μέλη, αλλά Υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι η απειλή ε, της γρήπης των πτηνών ή ε, επιδημίες ε, που μπορούμε καλύτερα να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Εκεί ανατρέπεται η αρχή της επικουρικότητας και η ίδια η αρχή της επικουρικότητας μας καλεί σε καλύτερο συντονισμό. Με τη βοήθεια μας λοιπόν και ε, την ε, υποστήριξη αυτό το θέμα ελήθη προς ικανοποίηση όλων. Τι κάνουμε για τον ιό ιτα 7 ή 9. Μέχρι σήμερα Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στις 2 Μαΐου έχει αναφέρει 128 ε, αποδεδειγμένα περιστατικά ε, σε άνθρωπο και όπως είπατε 26 ε, απεβίωσαν. Είμαστε σε στενή επαφή με τον ΠΟΗ ε, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς και Ελέγχου Νοσημάτων στη Στοχόλμη και είναι ένα πολύ εύγλωτο ε, παράδειγμα συντονισμένης απόκρισης και από την 31 31η Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κέντρο έχει κάνει δύο μελέτες αντικτύπου με τα κρατη πάντα και μια τρίτη τέτοια μελέτη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα η πηγή του ιού ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα και επίσης μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απόδειξη ότι μπορεί να μεταφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρόλο που στο μέλλον δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τέτοια μετάλλαξη. Και πάνω από 2.000 περιπτώσεις γρήπης ελέγχονται και δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο κίνδυνος διάδοσης της νόσου προς την Ευρώπη μέχρι σήμερα θεωρείται χαμηλός. Ωστόσο, οποιοδήποτε έχει ε, επιστρέψει από την Κίνα και δείχνει ε, σοβαρή αναπνευστική λίμωξη, ε, εξετάζεται, παρακολουθείται και έχουμε συμφωνήσει για μια ενδιάμεση μορφή ορισμού του ΙΤΑ 7 9 και όπως γνωρίζετε υπάρχει και μια επιτροπή για την ε, ασφάλεια υγείας ε, και για την έγκαιρη ε, προειδοποίηση και απόκριση. Και συνεδριάζουν, αύριο μάλιστα συνεδριάζει αυτό το δίκτυο. Και έχουμε και ένα μηχανισμό για να έχουμε και μία ανταλλαγή δειγμάτων, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να μπορούν να στείλουν στα εργαστήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάποια δείγματα, προκειμένου αυτά να αναλυθούν για να φανεί τελικά αν υπάρξει ιός. Μολονότι λοιπόν ο κίνδυνος ε, είναι χαμηλός, δεν επαναπαυόμαστε, Πρέπει να σας πω ότι πήγα πρόσφατα και στη μονάδα που έχουμε στο Λουξεμβούργο για να δω εκεί πέρα τι ακριβώς γίνεται για τις νόσους αυτές και πραγματικά μου έκανε εντύπωση τα όσα είδα εκεί, αλλά θα πρέπει πάλι να επαναπαυόμαστε. Ξέρετε ότι όλα τα πουλερικά τα οποία προέρχονται από την Κίνα αυτή τη στιγμή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι απάντησα στις, ε, σε όλες τις ερωτήσεις. Α, Σπαρτάμι, με συγχωρείτε. Ξέχασα να βρεθώ στην Σπαρτάμι. Έχουμε μία γνωμοδότηση από την Εύσα, η οποία το φθινόπωρο θα είναι έτοιμη. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμα από την Εύσα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρατηρήσεις, μάλλον ναι, πάρα πολλές συμβολές που έχει λάβει αυτή τη στιγμή η ΕΦΣΑ. Επομένως, ο ίδιος ο οργανισμός ζήτησε περισσότερο χρόνο για να καταφέρει να καταρτήσει την σφαιρική γνωμοδότησή της. Όσον αφορά τη βυσφενόλη α, όπως και όλες τις υπόλοιπε ουσίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία κοινή απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι δεν μας βοηθούν αυτή τη στιγμή οι εθνικές απαγορεύσεις. Περιμένουμε ακόμα να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της ΕΦΣΑ. Τώρα, όσον αφορά τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες, ε, ο κύριος Ποδότης είναι εκείνο αρμόδιος. Συνεργάζομαι πάντως με τη Γενική του Διεύθυνση και συμμετέχω στην όλη διαδικασία της επίπτωσης που μπορούν να έχουν ε, τα καλλιντικά στην ανθρώπινη υγεία. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια ενιαία κριτήρια για τους διαταράκτες αυτούς μέχρι τα τέλη του έτους. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. θα μπορούσαμε να προχωρούμε σε διάλογο μαζί σας και σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θέματα υπάρχουν πολλά, διότι υπάρχουν πολλά θέματα που απασχολούν και εσάς και εμάς. Ευχαριστώ εξ ονόματος των συναδέλφων μου για την συζήτηση και την απάντηση των ερωτήσεών μας. Μέχρι τέλους της εντολής μας θα έχουμε βέβαια ακόμα πολλές, πολλά πράγματα να κάνουμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάψει και αυτός ο κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι σωστό και σημαντικό αυτό που είπαν ορισμένοι συνάδελφοί μου, ότι είναι απαραίτητο ε, να συνδυαστούν, να συνδυαστεί, γιατί η οικονομία και η υγεία διασυνδέονται. Εμείς διεξάγουμε και συζήτηση μεταξύ των Προέδρων Επιτροπών, όπου εκφράζονται ιδέες και για μια διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρτοφυλάκια της Κομισιόν. Ε, αυτό ωστόσο με βρήκε εμένα κάθετα αντίθετο, διότι θέματα όπως υγεία και ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Πολύ ευχαρίστως σας βλέπουμε και θα σας ξαναδούμε. Η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται για τις 29 και 30 του μηνός, πάντα εδώ στις Βρυξέλλες. Σας εύχομαι καλή όρεξη και καλή επάνωδο για όσους επιστρέφετε.